and some silence is requested so that we may get started. Silence as we sit, take our seats, and thank you for that. Welcome everybody. Good afternoon. Καλώς ορίσατε. Καλό απόγευμα. Ξαναρχίζουμε λοιπόν, όπως το είχαμε συμφωνήσει, στις 3 ακριβώς, με το πολύ σημαντικό σημείο 7 Τη ημερησία διατάξεως που προβλέπει ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο κύριο Τζούλιαν Κίνγκ αρμόδιο για την Ένωση ασφάλεια Τον καλωσορίζουμε θερμά, θερμότατα μάλιστα θα πω. Ε, είναι πολύ ζεστή η μέρα αυτή στις Βρυξέλλες. Τι να κάνουμε, έχετε ε, στην, ε, στο φάκελό σας και αρμοδιότητες για την ασφάλεια και για ένα σωρό άλλα θέματα. Είχαμε την ευκαιρία ε, να έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Κίνγκ. Και είναι λοιπόν σημαντικό το γεγονό ότι η Επιτροπή μα ε, μπορεί ήδη να προβεί σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Κίνγκ τόσο νωρί, στο πλαίσιο δηλαδή τη νέα ε, θητεία του Κοινοβουλίου καθώς ε, η ασφάλεια αποτελεί βέβαια ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την Ευρώπη και φυσικά για τους πολίτες μας και αποτελεί ένα κατοχυρωμένο ε, θεμελιώδης δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πρόσφατα δημοσίευσε την 19η έκθεση προόδου της σε ό,τι αφορά την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και γνήσιας ένωσης ασφαλείας. Άρα λοιπόν αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον ε, την ενημέρωση από την πλευρά του Επιτρόπου Κίνξ σε ό,τι αφορά αυτή την 19η έκθεση, τη οποία σκοπό είναι να, να μα ενημερώσει ακριβώ σε σχέση με το τρομοκρατικό περιεχόμενο online, ε, την ε, στρατηγική εσωτερική ασφάλεια που συζητήθηκε και στο άτυπο συμβούλιο ΔΕΗ στο Ελσίνκι την περασμένη εβδομάδα και για τη διαλειτουργικότητα. Το ζήτημα της διαλειτουργικότητας ε, το συζητήσαμε διεξοδικά και αποτέλεσε δηλαδή ζήτημα που εντάσσεται μέσα στις αρμοδιότητες τη Επιτροπή μας σε ό,τι αφορά την διατηρητικότητα των μεγάλη κλίμακα συστημάτων πληροφορική ε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, τα σύνορα και τη μετανάστευση. Και εδώ βέβαια ε, μας απασχόλησε και το ζήτημα της ε, ε, επιβολής της νομοθεσίας και των υφιστάμενων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για να επιβάλλουμε ακριβώς την υφιστάμενη νομοθεσία. Η επιβολή της νομοθεσίας είναι πολύ σημαντική στον τομέα της ασφάλειας. Όταν έχουμε δηλαδή να κάνουμε με θέσπιση νέας νομοθεσίας, το πιο σημαντικό κομμάτι της είναι η σωστή επιβολή αυτής της νέας νομοθεσίας, των νέων εργαλείων. Και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε τον Επίτροπο King και τον ε, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα ακολουθήσουν. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τους συντονιστές ε, και μετά θα έχουν τη δυνατότητα και τα υπόλοιπα μέλη να πάρουν το λόγο. Να ε, σας υπενθυμίσω λοιπόν ότι πρώτοι θα πάρουν το λόγο οι συντονιστές μετά τον Επίτροπο. Παρακαλώ, Επίτροπε Κίνγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και βέβαια έχω αυτή τη δυνατότητα που σας συναντώ για πρώτη φορά εδώ στην Επιτροπή να σας πω ότι αναμένω με ενδιαφέρον την ε, συνεργασία μα. Βέβαια μια νέα λίμπε εδώ τώρα, με μια νέα σύνθεση, βλέπω κάποια νέα πρόσωπα και κάποια πρόσωπα τα οποία γνωρίζω και με τα οποία είχα τη δυνατότητα να συνεργαστώ στο παρελθόν. Ονομάζομαι λοιπόν Julian King, για ε, δεν έχω ξανασυναντήσει και ο, η δουλειά μου αν θέλετε είναι το να δημιουργήσουμε ε, με ισχυρότερη ένωση ασφάλεια. Αλλά πρωτού αναφερθώ λοιπόν στα ζητήματα τη πολιτική ασφάλεια, θα ήθελα να σα δώσω ένα γενικότερο πλαίσιο προς τα όσα προσπάθησα να κάνω κατά τελευταία χρόνια. Και ζητώ συγγνώμη από εκείνου οι οποίοι ήδη τα γνωρίζουν όλα αυτά. Θα αναφέρω λοιπόν αυτά τα βασικά ζητήματα και στη συνέχεια θα περάσω και στα βασικά θέματα που σας απασχολούν σε ό,τι αφορά τα εκκρεμή θέματα. Αποτελεί λοιπόν γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντιμετωπίσει κατά τελευταία χρόνια ε, πάρα πολλές απειλές ε, και κινδύνους. Ε, ξεκινώντας από την τρομοκρατία και ανέλαβα τα καθήκοντά μου το 2016 όταν είχαμε δηλαδή αντιμετωπίσει εκείνο το βήμα των φοβερών τρομοκρατικών επιθέσεων 15-16 ε, συνολικά σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ υπήρξε και ένα νέο κύμα κυβερνητικών απειλών αλλά και νέα είδη υβριδικών απειλών και επίσης αναδύθηκε σε αυτά τα χρόνια και ένα νέο είδος απειλής, δηλαδή η προστασία ε, για λόγους ασφαλείας της ε, κρίσιμες υποδομές μας. Για όλα λοιπόν αυτά τα ζητήματα, οι αρχές των κατώμελων παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η διασφάλιση δηλαδή ε, του να κρατούν τους πολίτες τους ασφαλείς. Σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα, είμαστε ισχυρότεροι εν τη όταν προσπαθούμε δηλαδή να τα διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Και αυτό ισχύει τόσο διεθνώ, όσο και ακόμα περισσότερο στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί λοιπόν από την πλευρά τη Επιτροπή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τη δουλειά μα, έτσι ώστε να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη ακριβώ προκειμένου να μα κρατούν ασφαλεί. Και αυτό το κάνουμε ε, με τη βοήθεια μια σειρά από εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μα μηχανισμού και μια σειρά από αρχέ, οι οποίε κάποιε από αυτέ είναι πολύ γνωστέ, όπω η Ευρωπόλ, ενώ υπάρχουν και άλλε οι οποίες δεν είναι τόσο γνωστέ, αλλά θα καταστούν πιο γνωστέ, όπω για παράδειγμα η νέα αρχή για την ε, ε, κύβερνο ασφάλεια. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και μια σειρά από διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότηση, ειδικότερα δηλαδή σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων μα στον τομέα τη ασφάλεια. Υπάρχουν επίσης και δίκτυα τα οποία κάποια από αυτά είναι πιο οργανωμένα ενώ κάποια άλλα είναι πιο άτυπα και όπου αυτό είναι απαραίτητο σε συνεργασία με εσάς θεσπίζουμε και νέα νομοθεσία και υπήρξαν δηλαδή μια σειρά από νομικές πράξεις οι οποίε ε, θεσπίστηκαν καν τα τελευταία χρόνια. Ξεκινήσαμε λοιπόν εστιάζοντα ιδιαίτερα στο ζήτημα τη τρομοκρατία, ακριβώ επειδή βιώναμε τότε εκείνο το ε, κύμα των ε, πολύ φρικτών τρομοκρατικών επιθέσεων το 2015 και 2016 πράγμα το οποίο έδωσε και ιδιαίτερη όθηση σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή το να δημιουργήσουμε μια πραγματική ένωση ασφάλεια στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναλάβαμε μία σειρά από πρωτοβουλίες έτσι ώστε να περιορίσουμε ε, τα πεδία εκείνα στα οποία έχουν δυνατόν να δραστηριοποιούνται οι τρομοκρατικές οργανώσεις και επίσης προσπαθήσαμε να ε, ενισχύσουμε την αντοχή μας, την, ε, την ισχύ μας απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις, αλλά και προσπαθήσαμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τον βίο εξτρεμισμό, είτε είναι τζιχαντικού τύπου, είτε για παράδειγμα ακροδεξιά, βία ή ακροδεξιά η οποία σε ορισμένε περιπτώσει αναλαμβάνει ακριβώ και τρομοκρατική δράση. Η ριζοσπαστικοποίηση λοιπόν σε αυτέ τι περιπτώσει λαμβάνει χώρα μέσα στι κοινότητέ μα, στι χώρε μα και ολόνα και περισσότερο λαμβάνει χώρα online, δηλαδή ειδικότερα μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Με την υποστήριξή σα λοιπόν, θεσπίσαμε κάποια μέτρα τα οποία καθιστούν πιο δύσκολη ε, τη μετακίνηση αλλά και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε πυροβόλα όπλα και σε κριτικά για του τρομοκράτε και ενισχύσαμε περισσότερο την ασφάλεια στα εξωτερικά μας σύνορα. Ενισχύσαμε ιδιαίτερα τις ε, αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της δημοκρατίας όπως η Ευρωπόλ ε, και επίσης ε, παρέχαμε και στοχευμένη χρηματοδότηση απέναντι σε πόλεις και οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την καλύτερη προστασία τους, χωρίς ωστόσο βέβαια να μεταβάλουμε τον επί αρχής ανοιχτό του χαρακτήρα. Επίσης ενισχύσαμε την κοινή μα αντοχή μέσω της ενίσχυσης των, ε, και της συνεργασίας ε, των συστημάτων επιβολής της νομοθεσίας μας. Και υπήρξαν μια σειρά από προτάσει ό,τι αφορά την διαλειτουργικότητα. Ένα ζήτημα δηλαδή που μα απασχόλησε και το οποίο συζητήσαμε επανειλημμένα με την προηγούμενη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ακριβώ προκειμένου να διασφαλίζουμε σε εκείνου που εργάζονται στην πρώτη γραμμή πρόσβαση στι απαραίτητε πληροφορίε, είτε πρόκειται για αστυνομικού υπαλλήλου, είτε για συνοριοφύλακε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά βέβαια η προληπτική δράση είναι πάντοτε καλύτερη από την εκ των υστέρων αντιμετώπιση. Έτσι λοιπόν προσπαθήσαμε τώρα να λάβουμε δράση και σε ό,τι αφορά την ριζοσπαστικοποίηση και ε, υπήρξαν μια σειρά από project από τα κάτω προς τα πάνω, όπου δηλαδή συμμετείχε και η κοινωνία των πολιτών ε, και οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς και δίκτυα όπως ε, το γνωστό σε πολλούς από εσά δίκτυο, δηλαδή το δίκτυο για την αντιμετώπιση της παστικοποίηση. Και επίσης λέμε κάποια μέτρα έτσι ώστε να ε, στοχεύσουμε πολύ ειδικά το τρομοκρατικό περιεχόμενο online. Ένα ζήτημα δηλαδή στο οποίο θα επανέλθω αργότερα στην ομιλία μου. Επειδή λοιπόν υπήρξε περισσότερη ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά την αναδυόμενη απειλή των ε, απειλών, ε, και των κυβερνοκινδύνο, αν θέλετε, κάναμε πιο πολλή δουλειά εδώ. Δηλαδή, προσπαθήσαμε καταρχήν να αναγνωρίσουμε τις απειλές εκείνες σε ό,τι αφορά την, τα δεδομένα μας και δημιουργήσαμε ακριβώς μια κοινή στρατηγική ασφαλεία σε σχέση με αυτές τι κυβερνοαπειλές, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την διεθνή συνεργασία, αλλά και ειδικότερα μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά και τον τομέα τη Άμυνα αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια εργαλειοθήκη, ένα toolbox σε ό,τι αφορά την κυβερνητική διπλωματία, έτσι ώστε να υπάρχει μια συντονισμένη αντιμετώπιση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιε απειλέ. Ε, και έχουμε προτείνει αποτρεπτικά μέτρα, για παράδειγμα, ε, ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία των αρχών επιβολή τη νομοθεσία, των διοκτικών αρχών. Από εκεί και μετά, εστιάσαμε στι απειλέ που βασίζονται ακριβώς στον κυβερνοχώρο, δηλαδή χρήση των δεδομένων τους ώστε να ε, επηρεαστεί η κοινή γνώμη. Και αυτό μας απασχόλησε, για παράδειγμα, ε, και στο πλαίσιο του τι μπορεί να συμβεί ε, προκειμένου να επηρεαστεί το αποτέλεσμα εκλογών. Και αυτό μας απασχόλησε και τώρα στο πλαίσιο των ευρωεκλογών. Και εδώ συνεργαστήκαμε και με την κοινωνία των πολιτών και τις δημόσιες αρχές, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε εκ των προτέρων να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα παραπληροφόρησης, προτού ξεκινήσει δηλαδή προεκλογική εκστρατεία, ε, των ευρωεκλογών και υπήρξε το σχετικό δίκτυο που ε, δημιουργήσαμε αλλά και ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης, ε, Rabbit Alert, έτσι ώστε να υπάρχει ταχεία ενημέρωση σε, σε σχέση με τέτοιου είδους προσπάθειες. Και επίσης κάτι που αποτέλεσε μια καινοτομία ήταν η συμφωνία από κοινού με τις, με τις πλατφόρμες μέσω κοινωνικής μια νέα στρατηγική σε ό,τι αφορά την διαχείριση τέτοιων δεδομένων, την αντιμετώπιση τέτοιων δεδομένων, μέσω της οποίας ακριβώς και σε συνεργασία με τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να έχουμε περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά αυτές τις πληροφορίες. με χαρά μου διαπίστωσα ότι δεν υπήρξαν και θα το διαπιστώσατε και εσείς ε, κάποιες ε, μεγάλου μεγέθους ε, επιθέσεις ή hacks ε, στο πλαίσιο των ευρωεκλογών, όπω για παράδειγμα είδαμε να συμβεί στις Ηνωμένε Πολιτείε ή για παράδειγμα κάποιε στοχευμένε επιθέσει ε, στο πλαίσιο τη ε, προεκλογική εξαρτησία του Πρόεδρου Μακρόν. Ε, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι στι ευρωεκλογέ δεν υπήρξε παραπληροφόρηση. Όχι, το αντίθετο ισχύει. Υπήρξε δηλαδή εκτεταμένη παραπληροφόρηση και ψευδεί ειδήσει και αναφέρθηκαν τέτοια φαινόμενα από την κοινωνία των πολιτών αλλά από και διάφορες αρχές και οι πηγές ήταν διάφορα bots, δηλαδή κάποιοι είτε πλαστοί λογαριασμοί είτε αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί, αυτά τα bots. Ε, και ε, αυτό δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε ως ε, τη νέα καθημερινότητα, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την, το πολιτικό γίγνεσθε. Θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και επίσης εξετάσαμε από εκεί και μετά το τι θα πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε έναν τομέα ο οποίος δυνητικά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ευάλωτο σημείο. Και αυτό αφορά τα πάντα, δηλαδή μέχρι και τις ζωές μας. Και αυτό είναι η υπεράσπιση της ψηφιακής μας υποδομής. Η συζήτηση εδώ, σε σχέση με αυτό το ζήτημα, εστιάζει ιδιαίτερα στο 5G. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν μία σειρά από περαιτέρω κρίσιμες τεχνολογίες ε, κρίσιμε υποδομέ τι οποίε θα ασφαλίσουμε. Σε ό,τι όμως αφορά το 5G, προτείναμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση του συστήματος που σημαίνει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να εντοπιστούν οι κοινέ απειλές και τα τροτά σημεία, τα ευάλωτα σημεία, έτσι ώστε να μειωθούν, να περιοριστούν αυτά τα ευάλωτα σημεία και έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια και έχουμε δεσμευτεί ότι μέχρι τα τέλη του έτου θα γίνει ακριβώ η ανάλυση των δυνητικών κινδύνων και των ευάλωτων σημείων, έτσι ώστε στο επόμενο βήμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ασφάλειά μα, είτε σε εθνικό επίπεδο τα κράτη-μέλη, είτε συλλογικά. Όμω ευθύ εξ αρχή είπαμε ότι ενδέχεται να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, του οποίου είναι πολύ δύσκολο και να περιορίσουμε και να διαχειριστούμε. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτή τη μελέτη που κάνουμε, τη ανάλυση ε, που κάνουμε και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτου, ίσω να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα προϊόντα, ορισμένε υπηρεσίε ή ορισμένη πάροχη υπηρεσιών να μην είναι ασφαλεί. Και από εκεί και μετά θα πρέπει να συζητήσουμε το τι σημαίνει αυτό, τι αντίκτυπο έχει. Όλη λοιπόν αυτή η δουλειά που κάνουμε, η οποία εντάσσεται ακριβώ στο πλαίσιο των εργασιών μα για την Ένωση Ασφαλείας, γίνεται πάντοτε λαμβάνοντα ιδιαίτερα υπόψη την προστασία των θεμελιωδιών δικαιωμάτων και ειδικότερα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, αυτό λοιπόν το ζήτημα βρίσκεται πραγματικά στην καρδιά ε, τη ε, πολιτική ασφαλεία μα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα στο παρελθόν και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και στο μέλλον. Εγώ πάντω ε, προσωπικά είμαι πεπισμένο ότι τα αποτελεσματικά μέτρα ασφαλεία θα πρέπει να βασίζονται και αυτό να είναι και προφανέ ότι βασίζονται δηλαδή στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γιατί στη διαφορετική περίπτωση τι ακριβώ προστατεύει αυτή η ασφάλεια, αν όχι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επίση, υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, Δικαστηρίου της Ένωσης δηλαδή, Εξετάσαμε τα εφιστάμενα μέτρα ασφαλεία στο πλαίσιο μια ε, έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε το 2015 και η οποία εξέταζε μέτρα ασφαλεία κατά τα τελευταία 10 πέντε χρόνια έτσι ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο πράγματι σέβονταν τα θεμελιώδη δικαιώματα και επίσης εξετάσαμε από εκεί και μετά περαιτέρω ε, νομοθεσίε όπω προέκυπταν νέα ζητήματα και νέε υποθέσει στο ε, δικαστήριο. Και επίση, ε, ήδη κατά την διατύπωση τη νέα μα πολιτική, δώσαμε ιδιαίτερο ρόλο και στην αρχή σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση. Δηλαδή είμαι περήφανο για το γεγονό ότι όταν κάναμε τι προτάσει μα για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεγάλη κλίμακα, συμπεριλάβαμε το EDPS και το FRA δηλαδή αυτές τις αρχές ακριβώς σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Βέβαια, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πάντοτε τα πάντα σωστά. Ε, όχι. Ε, οι αρχικές μας προτάσεις δεν είναι πάντοτε ολόσωστες και γι' αυτό ακριβώς είναι απαραίτητο ο διάλογος ο οποίος γίνεται και με εσά ε, και ο οποίος θα συνεχίσει να λαμβάνει η χώρα. Έτσι ώστε δηλαδή να ελέγχονται αυτές οι προτάσεις της Επιτροπής από εσάς και να ελέγχονται διεξοδικά. Έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κατά την οικοδόμηση της κοινή μας ασφάλειας δεν υπονοβεύουμε κανέναν τρόπο τις, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αξίες μας. Όπως είπε ο Πρόεδρος, ορισμένα από αυτά τα ζητήματα αναφέρονται και μέσα στην 19η έκθεση πρόοδου σε ό,τι αφορά την Ένωση Ασφαλεία. Εκεί λοιπόν στην έκθεση αναφέρονται οι περαιτέρω εκκρεμότητε, αν θέλετε, των οποίων θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού. Ε, και υπάρχουν και κάποιε νομικέ πράξει, νομικέ προτάσει, επί των οποίων ε, ελπίζω πω θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο μέσα στου ε, επόμενου μήνε. Και υπάρχουν και κάποια περαιτέρω ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω μέχρι τα τέλη του έτους. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση, θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε την έκθεση ω προ το τι ακριβώ συνέβη στο πλαίσιο των ευρωεκλογών και από εκεί και μετά θα πρέπει να εξετάσουμε και τι πρακτικέ ε, που εφαρμόζονται από τι ε, πλατφόρμες των μέσων κοινωνική δικτύωση. Και με βάση αυτέ τι εκθέσει ενδεχομένω να χρειαστεί να θέσουμε κάποιε προτεραιότητε ακόμα και αν αυτές οι προτεραιότητες ετευθούν από τη Νέα Επιτροπή. Επίση, θα χρειαστεί να ε, εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα του 5G και των κρίσιμων υποδομών μα. Ε, όπω είπαμε, σχετική ανάλυση που γίνεται θα τρέξει μέχρι τα τέλη αυτού του έτου. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα επί των οποίων θα ήθελα να προβούμε σε ένα διάλογο στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα εκρεμή νομοθετικά ζητήματα. Υπάρχει μία δέσμη προτάσεων, όπω θα γνωρίζετε, που έχει τεθεί επιτάπητο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τρομοκρατικού περιεχομένου online. Αναφέρθηκα σε αυτό το ζήτημα λίγο προηγουμένω ε, πρωτήτερα στην ομιλία μου. Δηλαδή, αυτό το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο εξακολουθεί να παραμένει online σε μεγάλο όγκο. Δηλαδή, κατά τα τέλη ε, του περασμένου έτους, παρότι το ΆΣΕΣ είχε διαλυθεί ουσιαστικά, το τρομοκρατικό περιεχόμενο που ε, σχετίζεται με αυτούς είχε πραγματικά αυξηθεί και είχε φτάσει στα επίπεδα του 2015. Άρα λοιπόν υπάρχει υπερβολικά μεγάλος όγκος τέτοιου τρομοκρατικού περιεχομένου και μάλιστα περιεχομένου το οποίο είχε εντοπιστεί στο παρελθόν και δεν είχε ακόμα απομακρυνθεί, ενώ παρουσιάζονται λόγω και περισσότερε πλατφόρμε. Σε μια μελέτη, για παράδειγμα, που έγινε από αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε τέτοιου είδου παράνομο, παράνομο εξτρεμιστικό, τσιγχατιστικό περιεχόμενο σε περισσότερε από 400 πλατφόρμες. Γι' αυτόν ακριβώ το λόγο προτείνουμε ακριβώ να βασιστούμε στην προαιρετική, την εθελοντική συνεργασία, πολύ αποτελεσματική που είχαμε ε, και στο παρελθόν, ειδικότερα με τις μεγάλες κλίμακες ε, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά από εκεί και μετά αυτά ε, δεν είναι αρκετά και δεν κινούνται και αρκετά γρήγορα. Και φυσικά με τέτοιου είδους μέτρα δεν καλύπτουμε και τον απαραίτητο αριθμό των πλατφορμών που θέλουμε. Γι' αυτό λοιπόν, όπως γνωρίζετε, πέρσι υποβάλαμε μια πρόταση η οποία καθιστά υποχρεωτική την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου μετά από τη λήψη μια τέτοια εντολή αφαίρεση του περιεχομένου από μια αστυνομική δικαστική αρχή. Και επίση αυτή την πρόταση ε, προβλέπεται ότι αν μια πλατφόρμα ε, χρησιμοποιείται συστηματικά για την διάδοση τέτοιου είδου τρομοκρατικού περιεχομένου, θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση με τι αρμόδιε αρχέ ω προ το ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει η χρήση τη για αυτού του σκοπού. Και εκείνο που είναι ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δεσμεύσουν, να αφιερώσουν δηλαδή συγκεκριμένε ικανότητε από τι διοκτικέ του αρχέ και του απαραίτητου πόρου για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματο. Άρα λοιπόν, παρότι αυτό ήδη συμβαίνει, προτείναμε πλέον να, είναι, να αποτελεί δεσμευτική υποχρεωτική διάταξη. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε πως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά αυτό το περιεχόμενο. Ε, και φυσικά υπάρχει και το δικαίωμα τον, ε, υπάρχουν τα έντικα μέσα σε περίπτωση που κάποιος θεωρεί, θεωρήσει πως ε, είναι άδικο κάτι τέτοιο. Και αυτή η προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της ε, διεθνής προσπάθειας που γίνεται για παράδειγμα στο, στο επίπεδο των συζητήσεων του G7 ή για παράδειγμα σε συνέχεια της δημοκρατικής επίθεσης που έγινε στη Νέα Ζηλανδία και τη συζήτηση που ακολούθησε. Και βέβαια αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα κάνουμε μαζί σας αυτό το θέμα το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να φτάσει ε, σε μια ε, συμφωνία σε ό,τι αφορά την πρώτη ανάγνωση σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Οπότε θα δούμε, Πρόεδρε, σε ποιο βαθμό θα είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία το ταχύτερο δυνατό σε σχέση με το τρομοκρατικό περιεχόμενο. Επίσης, η βελτίωση της πρόσβασης των διοκτικών αρχών στα, ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία παραμένει ένα ακόμα ζήτημα που θα μας απασχολήσει. Και είναι ένα ε, μεγάλο πρόβλημα γιατί οι μισές από τις ε, ποινικέ ε, έρευνες σε σχέση με δηλαδή, δικαστικές υποθέσεις που εξετάζονται σήμερα έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε άλλη δικαιοδοσία, σε άλλο κράτος μέλος και οι σχετικές διαδικασίες είναι πολύ αργές και διοικητικά επαχθείς και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε πολλές υποθέσεις οι οποίες τελικά δεν καταλήγουν έτσι όπως πρέπει ακριβώς επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία και θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, η πρόταση λοιπόν την οποία υποβάλαμε συζητήθηκε ε, μακρόν από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Αντιλαμβανόμαστε πως τα ζητήματα που θέτουμε εκεί είναι δύσκολα, αλλά ελπίζω πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο και να προχωρήσουμε. κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι το ότι θα πρέπει να κάνουμε μια πιο εκτενή συζήτηση ε, σε σχέση με, και με την προηγούμενη έκθεση ΤΕΡ που είχε συνταχθεί κάτι του προηγούμενου κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το τι θα πρέπει να κάνουμε σε σχέση με τους ε, τρομοκράτες ε, μαχητές και τις οικογένειάς τους γιατί κάποιοι ήδη ακόμα βρίσκονται σε ζώνες ένοπλης σύραξη στο Ιράκ και στη Συρία. Και οι αριθμοί εδώ μας εκπλήσουν γιατί Γύρω στους 5.500 ε, ξένοι μαχητές έχουν καταλήψει τις χώρες μας προκειμένου να μεταβούν σε αυτές τις ε, εμπόλμες ε, ζώνες, στο Ιράκ δηλαδή και στη Συρία. Και τα τρία τέταρτα αυτών ήταν άνδρες, ενώ γύρω στο ένα τέταρτο ήταν γυναίκες. Και φυσικά εδώ δεν είναι ακριβή αυτά τα νούμερα, αλλά γύρω στους 1.400 μαχητές έχασαν τη ζωή τους και ίσως αυτός ο αριθμός να είναι και ψηλότερο. και επί τη βάση των όσων μας έχουν διαβιβάσει ως πληροφορίες τα κράτη-μέλη γύρω στα 1600 άτομα αυτοί οι μαχητές δηλαδή που εγκατέλειψαν τις χώρες τους έχουν επιστρέψει ήδη. Ε, ε, ειδικότερα δηλαδή εκείνοι του πρώτου βήματος, ε, του πρώτου κύματος συγγνώμη, που αποχώρησαν. Άρα έχουμε γύρω στις 3.000 οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχουν απογίνει δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Βρίσκονται στις, στο Ιράκ και στη Συρία. Βρίσκονται σε, σε άλλες ε, ένοπλες όπου θεωρούν δηλαδή ότι θα πρέπει να ε, αγωνιστούν. Πάντως γνωρίζουμε ότι γύρω στου 600 ε, άντρε και γυναίκε και γύρω στα 700 παιδιά βρίσκονται υποκράτηση. Το μεγαλύτερο μέρος τους στη Συρία. Σε περιοχές δηλαδή ελεγχόμενες από Κούρδους της Συρίας. Και θεωρούμε πως γενικά στην περιοχή υπάρχουν 1.400 παιδιά, εκ των οποίων ε, ένας από τους δύο γονείς έχει ε, κατά τους μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ε, το κατά πόσο θα πρέπει να επαναπατρίζονται τέτοιου είδους άτομα, τέτοιου είδους μαχητές, αποτελεί ένα ζήτημα από το οποίο αποφασίζουν τα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχουν εδώ πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε από κοινού για να παράσχουμε βοήθεια. Έχουμε δηλαδή συζητήσει ήδη το ζήτημα της παροχής υποστήριξης σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ε, δίωξη των μαχητών που επιστρέφουν στις χώρες τους ε, και σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό τους σε αυτές τις περιοχές αλλά και σε άλλες γειτονικέ χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν ένα αντίστοιχο πρόβλημα και επίσης μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω το πώς ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των παιδιών. Πρόκειται λοιπόν εδώ ε, για δουλειά την οποία θα πρέπει να κάνουμε και στο μέλλον. Και άλλε προτάσει τη Επιτροπή ε, ΤΕΡ για την τρομοκρατία έχουν ε, τεθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό έγκλημα. Αλλά το τελευταίο που ήθελα επίση να αναφέρω, ευχαριστώ που μου δώσατε τόσο χρόνο, είναι ότι όπω είπε και ο πρόεδρος στην αρχή, το θέμα δεν είναι μόνο να κάνουμε καινούργια πράγματα, είναι να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε και σωστά αυτά τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει. Και σε αυτό το τομέα ίσως περισσότερο από άλλους τομείς πολιτικής, η εφαρμογή, εφαρμογή, εφαρμογή πρέπει να είναι το κύριο καθήκον μας. Και σας διαβεβαιώ ότι συνεργαζόμενος ε, με εσά θα προσπαθήσω να υλοποιήσω αυτά που αποφασίσαμε μαζί, είτε είναι νομοθεσία, βοήθεια για τους ε, διάφορους ενωσιακούς φορείς, ε, στήριξη για τα, δίκτυά μας. Όλα αυτά πρέπει να μπορέσουν να, να, μπορέσουν να λειτουργήσουν. Η τελευταία έκθεση λοιπόν προόδου Μα λέει τι γίνεται για την εφαρμογή των βασικών νομοθετικών κειμένων στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον όσο θα έχω αυτή τη θέση, θα συνεχίσω να αξιοποιώ κάθε δυνατότητα που έχουμε για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, αλλά επίση για να ε, καταδείξω τις ευθύνες τους εάν υπάρξουν παραβιάσεις ή ανεπάρκειες. Καταλήγοντας, νομίζω ότι κάναμε μαζί ε, χρήσιμα πράγματα κατά την τελευταία θητεία. Πολλά ακόμη πρέπει να κάνουμε. Οι απειλέ αυτέ συνεχίζουν να εξελίσσονται, να μεταβάλλονται. Πρέπει λοιπόν και εμεί να ε, προσαρμοζόμεθα. Και προσβλέπω στην πολύ στενή συνεργασία με τη νέα σα επιτροπή του επόμενου μήνε και σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που και πάλι επιδείξατε την ε, πολιτική σας βούληση για να ανταλλάσσετε τακτικά απόψεις με την Επιτροπή μας, όπως κάνατε και πριν τις εκλογές. Σωστά υπενθυμίσατε τη συνόψιση του πλαισίου. Έχουμε τις προηγούμενες εκθέσεις, αλλά κυρίως Πώ είχαν τα πράγματα το 14, 15, 16 που είχαμε τι διάφορε τρομοκρατικέ επιθέσει, σοβαρότατου κινδύνου, επιθέσει που εκδηλώθηκαν ε, στο μήκο και το πλάτο τη Ένωση, οπότε συνειδητοποίησαμε ότι χρειάζεται μια ενωσιακή ανταπόκριση, αντίδραση, περισσότερο παρά ποτέ. Συνοψίσαμε την έκθεση που είναι στη διάθεση των μελών τη Επιτροπή. Και αναφερθήκατε και σε κάποια άλλα στοιχεία της έκθεση αυτής που πρέπει να συζητηθούν σωστά τους επόμενους μήνες. Για παράδειγμα αυτοί οι ξένοι μαχητές. Η Επιτροπή της Europol που δημιουργήθηκε μετά από αίτημα της ΛΥΜΠΕ και η παρακολούθηση των θεμάτων ε, κυβερνοασφάλειας από την Επιτροπή μας καθώς επίσης και κάποιου είδους παρουσία της Επιτροπής μας στις ε, διυπουργικές ε, συνεδριάσεις του φόρουμ για το ίντερνετ. Η επόμενη συνεδρίαση είναι τον Οκτώβριο, μέσα Οκτωβρίου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε αυτό μας το αίτημα μετά τις διακοπές. Τώρα παρακαλώ οι συντονιστές Παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένα γιατί έχουμε πίεση χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει επαρκή χρόνο και για του υπόλοιπου συναδέλφου γιατί έχω εδώ ένα κατάλογο με πολλά ονόματα και βλέπω και άλλοι τώρα να εκδηλώνουν την ε, επιθυμία τους. Λοιπόν, παρακαλώ κύριοι και κυρίες και κύριοι συντονιστές, δύο λεπτά για να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε ερωτήσεις στον Επίτροπο Κίν και για να έχει χρόνο βεβαίως να απαντήσει. Λοιπόν, ΕΛΚ. Εσείς εκπροσωπείτε το ΕΛΚΑ. Α, α εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε Κίνγκ, λέει ο κύριος Λέναρς, που είστε εδώ στην αρχή της αιτίας μας. Η ασφάλεια ήταν ε, μεγάλη προτεραιότητα την τελευταία πενταετία για την Ένωση και θα συνεχίσει και την επόμενη πενταετία. Και ως ΕΛΚΑ ε, προσβλέπουμε στην περαιτέρω στενή συνεργασία μαζί σας. Λοιπόν, ταχαίως. ηλεκτρονικά στοιχεία και την ε, συνεχιζόμενη εργασία στο νομοθετικό πακέτο, αλλά το Συμβούλιο επίσης ενέκρινε την ε, διαπραγματευτική εντολή για την διάσκεψη για της Βουδαπέστης και για τη Συμφωνία Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε χρονοδιάγραμμα για αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και πώς θα διασφαλίσετε ότι ότι αποφασιστεί για αυτά τα δύο θέματα θα συμφωνεί με αυτά που περιέχονται στο δικό μας νομοθετικό πακέτο χωρίς παρόλα αυτά να καθυστερήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Για το PNR, στη συνάντηση Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών σε υπουργικό επίπεδο συμφώνησαν δύο πλευρές να γίνει μια αξιολόγηση της συμφωνίας των δύο μερών για το PNR στην ανακοίνωση τύπου υπόθηκε ότι θα αξιολογηθεί η τρέχουσα συμφωνία. Θα αξιολογηθεί επίσης και το επίπεδο των προδιαγραφών που έθεσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, στην απόφασή του για τη συμφωνία με τον Καναδά και πώς θα προσαρμοστεί τότε λοιπόν και η διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ. Και μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για την εφαρμογή του PNR στα κράτη-μέλη. Διαλειτουργικότητα το είπατε. Πολλά κάναμε γι' αυτό ως σώμα μαζί με εσά, ούτω ώστε να εγκριθεί αυτό το πακέτο πριν την προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα περνάμε στην εφαρμογή. Όπως είπατε, δεν τα πάμε πάντα πολύ καλά στην εφαρμογή, άρα πρέπει στενά να παρακολουθείτε και με στιβαρό χέρι την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας. Μπορείτε να μας ενημερώσετε λίγα για το πώ πάει αυτό το θέμα. Τέλος. Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Βεβαίως θα ξεκινήσουν οι τριμερείς διάλογοι. Αλλά αυτό αφορά μόνο τη δική μας επικράτεια. Αναφερθήκατε σε αυτά που έγιναν στην Νέα Ζηλανδία, στο Christchurch και την έκκληση που υπάρχει. Ε, δεν ε, περιέχονται όμως αυτά που λέγονται, ε, δεν περιέχουν τις ΗΠΑ και πολλές από τις 400 πλατφόρμες. Τι μπορούμε να κάνουμε διμερώς με τις ΗΠΑ για να διασφαλίσουμε ότι το τρομοκρατικό περιεχόμενο που πρέπει να απαλήφεται, να απαλήφεται. Συγγνώμη, μίλησα λίγο παραπάνω. cards were also raised, so I... Λοιπόν, Κοιτάξτε, θα χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένας. Η κυρία Ζίπελ. Ναι, αλλά Πώς να μιλήσω τόσο σύντομα, πολλά θέματα ανέφερε ο Επίτροπος. Πρώτα απ' όλα, σήμερα το πρωί και για ένα εντελώ διαφορετικό θέμα αναφερθήκαμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Πολύ συχνά υπάρχει ευρεία συνένεση για ένα νέο νομοθέτημα, αλλά μετά κολλάμε στην εφαρμογή για τον ποινικό κώδικα και την ε, ανασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλούς νόμους αλλά όταν συζητάμε με τους αστυνομικούς και τους δικαστικούς, μας λένε, μα δεν έχουμε ούτε χρόνο, ούτε πόρους, ούτε προσωπικό, ούτε εξοπλισμό για να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Όλα αυτά που αποφασίσατε εσείς. Να τα εφαρμόσουμε, όχι να τα βλέπουμε γραμμένα. Ποια είναι η δική σας ε, άποψη για το πώς τα πάνε τα κράτη-μέλη. Επίσης λέμε πολλά για την τρομοκρατία και την εξτρεμιστική βία. Και σας ευχαριστώ που αναφέρ, αναφερθήκατε στην ανάγκη να υπάρξει και πρόληψη. Αλλά σε διάφορα μέρη της Ένωσης ε, και στη Γερμανία, αλλά τώρα πρόσφατα και στην Πολωνία, διάφορες χώρες λοιπόν, έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που λείπει είναι πολιτική βούληση για να καταπολεμήσουμε τον βίο εξτρεμισμό και την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων κάποιων ομάδων συμπολιτών μας. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό, κάνουν αρκετά τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση του βίου εξτρεμισμού. Επίσης είπατε ότι όσα κάνουμε για τον ποινικό νόμο και την ασφάλεια πρέπει να γίνονται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε μεμονωμένε οδηγίες, να βλέπουμε και το δάσο. Εάν ε, ένα ε, μέτρο αποδυναμώνει θεμελιώδη δικαιώματα στον α τομέα και ένα άλλο μέτρο αποδυναμώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα σε άλλο τομέα, πρέπει να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση. Είναι όντω σεβαστά γενικά μέσω τη όλη πανοπλία των μέτρων που ε, υιοθετούμε. Διασφαλίζουμε την εφαρμογή του. Έχουμε μια τέτοια σφαιρική επισκόπηση. Αν υπάρχει, πείτε μου πού μπορώ να τη βρω. Και τώρα αυτό που λέτε για τα ηλεκτρονικά στοιχεία Κοιτάξτε, δεν είναι στοιχεία. Καλύτερος, ε, καλύτερος όρος θα ήταν να λέμε για ηλεκτρονικά κείμενα, πράγματα. Αν θα γίνουν στοιχεία μιας ε, δικαστικής έρευνας θα φανεί αργότερα. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά με τους κοιόδης για τα θέματα αυτά τους τελευταίους μήνες και ευχαριστώ για την συμμετοχή τους και υπάρχουν ανησυχίες για διάφορους ε, τομείς και καλό είναι που τα συζητάμε όλα τα προβλήματα και ελπίζω ότι τώρα μπορούμε να, αρχίζουμε, να αρχίσουμε να υποβάλουμε τα αιτήματά μας μέσω τροπολογιών. Γιατί πραγματικά πρέπει να σεβόμεθα, ε, με μεγάλη προσοχή τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πραγματικά πρέπει να επιμείνω, λέει ο Πρόεδρος, να μην ξεπερνάτε τα δύο λεπτά, γιατί διαφορετικά, όπως είπα και προηγουμένως χαριτολογώντας, θα χρειαστούμε και μεγαλύτερη βάρκα. Uh, Κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, ε, ελπίζω ότι και τα αποτελέσματα θα είναι τέτοια που θα σας έχουμε κοντά μας για πολλά χρόνια ακόμα. η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολύ καλά μερικά πράγματα, δηλαδή να κάνει νόμους. Ε, αυτό μπορεί να είναι ελκυστικό και εδώ ερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, τις, ε, ε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και λέμε τι ωραία που τα κάναμε και περάσαμε και αυτή την νομοθεσία. Το θέμα είναι όμως και η αξιολόγηση και η υλοποίηση εκεί. Πραγματικά έχουμε πολύ κακές επιδόσεις, πολύ κακές επιδόσεις και αν δείτε και το, την, τον πίνακα επιδόσεων όσον αφορά ένα σωρό ζητήματα, ε, ας πούμε τέσσερα χρόνια μετά από την τελική προθεσμία. Η οδηγία για το ξέπλυμα του χρήματος ακόμα σε 24 χώρες μέλη δεν έχει ενσωματωθεί. Ε, σε 24 χώρες πώς είναι δυνατόν αυτό. Η αξιολόγηση επίσης το ίδιο. Ε, στην ουσία καλούμαστε να αξιολογήσουμε την επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Και αυτό το κάναμε ήδη ήδη από το 2011 και ακόμα περιμένουμε την πρακτική εφαρμογή. Το PNR που ακούστηκε προηγουμένως, ε, το Bundeskriminalakt στη Γερμανία ε, απεφάνθη ότι ε, με το PNR 99,7% των ετοιμάτων τελικά βγαίνουν θετικά και η Κομισιόν λέει «Α, αυτό όμως δεν είναι καλό για και σε σχέση και με όλα τα συστήματα για τα ε, δεδομένα. Ωραία. Λέτε ότι λαμβάνουμε υπόψη πάντοτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα κτλ. Πολύ ωραία. Αλλά πόσοι είναι αυτοί οι νόμοι που ε, στην ουσία εμείς τι καταψήφιμε, αλλά δεν έχει σημασία, ε, τελικά ε, απορρίπτονται από, από το δικαστήριο, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αναλογιστείτε λίγο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι νομικός ορθή, ορθά τα νομικά μας κείμενα και η νομοθεσία μας. Εν πάση περιπτώσει πιστεύω ότι ναι, πραγματικά πρέπει να καταπολεμήσουμε την ε, τρομοκρατία κτλ. Αλλά να μην ε, κλείνουμε και τα μάτια προς την, ε, τον ακροδεξιό εξτρεμισμό. Υπάρχει ε, βία όχι μονάχα και από τις εγκληματικές οργανώσεις αλλά και από κάποιους ε, πολιτικούς ε, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα διαρκώς σε ομοφιλόφιλους κλπ. Λοιπόν, όταν λέω ότι μερικές φορές μπορεί να είναι νόμιμο το περιεχόμενο αλλά πολύ συχνά μπορεί και να μην είναι σωστό. Η κυρία Σκρίκτα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Κίνγκ για την εργασία του όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κυβερνοεκκλήματος καθώς επίσης ε, και για το ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει με σύγχρονο τρόπο τις εξελίξεις ε, στο, στο, στο σε αυτούς πράγμα όχι πάρα πολύ ε, εύκολο. Βεβαίως δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τις βασικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου Οποιαδήποτε κίνηση γίνεται για καταπολέμηση εγκλήματο, τρομοκρατία κλπ. δεν θα πρέπει να υπονομεύει από την άλλη πλευρά αυτές τις αξίες και τις αρχές. Έχω δύο συγκεκριμένε ερωτήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό ενισχύουμε διαρκώς τις αρχές της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας. Αλλά αναρωτιέμαι, βλέπετε να υπάρχει ανάγκη ε, για μεγαλύτερη διασφάλιση των ε, δικαιωμάτων στις διαδικασίες ας πούμε που εμπλέκουν υπόπτους κλπ. Ε, υπάρχουν βεβαίως ε, μεγάλες διαφορές όσον αφορά ε, τα θέματα αυτά μεταξύ των κρατών μελών παρότι υπάρχει και το σύστημα της δικαστικής αρρωγής. Επομένως άνθρωποι που χρειάζονται διασφαλίσεις και διασφάλιση και των δικαιωμάτων και δικλείδες ασφαλείας αυτό πρέπει να το δείτε λίγο. Κάτι άλλο, πιλωτικό πρόγραμμα για την αναθεώρηση του συστήματος και των προγραμμάτων συλλογής δεδομένων ε, αυτό έχει αρχίσει και λειτουργεί εδώ και κάποια χρόνια. ρωτιόμαστε μήπως η Κομισιόν είναι σε θέση πλέον να ε, μας πει ποια είναι τα ευρήματα και ποια είναι τελικά η αξιολόγηση που μπορεί να κάνει για αυτό το πιλωτικό. Ε, πρόγραμμα γιατί μπορεί να προκύψουν νέα προγράμματα, νέες προτάσεις ε, που θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο την διακράτηση των ε, δεδομένων. Αναρωτιέμαι λοιπόν κύριε Κίνγκ, κατά την άποψή σας είναι απαραίτητο και ανάλογο να διευρύνεται ακόμα περισσότερο τα συστήματα και το χρόνο διακράτησης των στοιχείων μη Μήπως ε, μπορείτε να μας πείτε κάτι και την προσωπική σας άποψη όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Καρντίνο και μετά ε, ε, ο κ. Προκατσίνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Επίτροπο γιατί είναι σήμερα εδώ, καθώς επίσης και γιατί δημοσίευσε και την έκθεση για την 19η έρευνα βεβαίως. Όταν θα δημοσιευτεί κανονικά θα την διαβάσουμε και θα την αξιολογήσουμε δεόντως. Πιστεύουμε πάντως ότι οι προκλήσεις και οι απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουμε είναι όλο και πιο περίπλοκες και επομένως θα πρέπει με ακόμα καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια, το θέμα της ασφάλειας των πολιτών μας. Οργανωμένο έγκλημα, ε, ε, έγκλημα ε, και τρομοκρατία. Είπατε ότι κύριο μέλημα είναι να είναι ασφαλείς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Άρα θα πρέπει να δούμε λίγο και το θέμα της ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα. Η Ιταλία βρίσκεται στο, στην πρώτη γραμμή του μετόπου θα πρέπει να βοηθηθεί. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε με ε, ε, ρόμη και στιβαρότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Πρώτη ερώτηση λοιπόν, ποια είναι τα μέτρα, τα αποτελεσματικά τα οποία μπορούμε να ή μπορείτε να προβλέψετε για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων. Βεβαίως εδώ υπάρχει και ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα που είναι το trafficking. Δεύτερη ερώτηση, όσον αφορά την καταπολέμηση του trafficking, με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, διασφαλίσει την σωστή εφαρμογή της οδηγίας αντιτράφικινγκ. Ε, Επίσης, ε, η Κομισιόν προτίθεται να λάβει υπόψη ε, το σουηδικό ε, μοντέλο όπου στην ουσία ένοχος θεωρείται αυτός ο οποίος παίρνει τις, λαμβάνει τις υπηρεσίες, τις εξωτερικές υπηρεσίες και όχι αυτός που τις προσφέρει που είναι θύμα. Ευχαριστώ πολύ. Προκατσίνη. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που είστε σήμερα εδώ πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι η Κομισιόν πρέπει να ασχοληθεί και με τη διαδικασία ρίζοσπαστικοποίησης ε, που ε, στην ουσία διαμορφώνει αυτούς τους τρομοκράτες ε, από τους οποίους πρέπει να αμυνθούμε. Δεν έχει γίνει κάποια ανάλυση για το πόσοι από αυτούς τους ενεργούς στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια ε, τρομοκράτες έχουν διαμορφώσει την ε, δράση τους ας πούμε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή είναι από από αυτούς που έχουν έρθει με τα τελευταία μεταναστευτικά κύματα. Είπατε ότι τα κράτη-μέλη έχουν κυριαρχία όσον αφορά την όσον αφορά την ε, ασφάλεια, αλλά μονάχα ε, οι κοινέ ε, απειλέ είναι αυτέ που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η άποψή σα όμω για αυτέ τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που συστηματικά παραβιάζουν την κυριαρχία μα. Η Κορνίλια Χέρνστε δεν είναι εδώ από την Γκουε. Θέλει κάποιος άλλος από την ΚΟΕ να πάρει το λόγο. Όχι από ό,τι φαίνεται. Προτείνω λοιπόν να ανοίξουμε ε, να έχουμε ένα πρώτο γύρο απαντήσεων μετά από τις ερωτήσεις των συντονιστών και μετά να ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ θερμά όλους όσους ε, παρακολουθούν αυτά τα ζητήματα εδώ και κάποιο καιρό και γι' αυτό ε, γρήγορα στις λεπτομέρειες που είναι και σημαντικές. Δεν ναι, θα ακολουθήσω τη σειρά με την οποία τέσαν ερωτήσεις και ελπίζω να μην ε, ξεχάσω καμία από αυτές. Να πω ότι υπήρξαν μία σειρά από ερωτήσεις σε σχέση με τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, το e-evidence. Ε, και ίσως θα πρέπει να μιλήσετε και με την Επίτροπο Βεραγιουρόβα αύριο, την οποία θα συναντήσετε δηλαδή εδώ αύριο στην Επιτροπή, ε, θα πρέπει λοιπόν να τη ρωτήσετε και εκείνη για αυτό το ζήτημα. Ε, εμείς θα συνεχίσουμε να το προωθούμε από κοινού και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά α, ε, τους περιορισμούς που μας θέτει το χρονοδιάγραμμά μας γιατί έχουμε συμφωνήσει από αυτή τη εντολή και το κάναμε επειδή ε, όπως θα σας πει και αύριο πιο δεξιοδικά η Βέρα ε, έχουμε ξεκινήσει το διάλογο με τι Ηνωμένε Πολιτείε, γνωρίζοντας βέβαια ότι ο διάλογο παραμένει ανοιχτό και ακόμα υπάρχει ε, ε, μέλλον σε σχέση με αυτόν τον ε, διάλογο και σε ό,τι αφορά και την δική μα ε, θέση, την οριστικοποίηση τη θέση μα. Και αυτό γιατί οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται πιο μπροστά από εμά σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Έχουν δηλαδή το Cloud Act και ήδη έχουν κινήσει και διμερεί. ε, ε επαφές με κάποια κράτη-μέλη έτσι ώστε να υποστηρίξουν τη δική τους ε, προσέγγιση η οποία ακριβώς ε, στοχεύει περισσότερο στη σύναψη διμερών συμφωνιών και όχι στη σύναψη μιας συμφωνίας με το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατά τη δική μου άποψη θα μπορούσε να έχει για ισχυρότερες και πιο αξιόπιστες δικλείδες ασφαλείας. Αν αλλά ήδη στην πρόταση που έχει υποβληθεί σε σχέση με μια τέτοια συλλογική ε, πρόταση υπάρχουν πράγματι πιο ισχυρέ δικλείδε ασφαλεία. Άρα λοιπόν ε, η Βέρα θέλει να προωθήσει αυτό το διάλογο. Τώρα σε ό,τι αφορά ε, το Συμβούλιο τη Ευρώπη και τη διαδικασία τη Βουδαπέστης. Εμεί θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το διάλογο και ο επόμενο γύρο συζήτηση θα κινηθεί το Σεπτέμβριο. Οπότε εμεί θέλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά εκεί στον Λόγο φόρουμ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνδιαμορφώσουμε την ε, συζήτηση αυτή, καθώ σε αυτήν περιλαμβάνονται και μία σειρά από τρίτε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών θα διασφαλίσουμε ή θα, θα φροντίσουμε μάλλον το ότι τα όσα λέμε ε, προς τα έξω τα απηχούν τα όσα ακριβώς συζητούμε εμείς εδώ και τα όσα δεσμεύουμε και θα βρισκόμαστε σε επαφή και αν ε, φυσικά εσείς θα έχετε την ε, αίσθηση ότι κάτι, κάτι κάνουμε λάθος σίγουρα θα μας το αναφέρετε. Τώρα, τέθηκαν μια σειρά από ερωτήματα σε ό,τι αφορά την οδηγία PNR. για τις καταστάσεις των επιβατών. Έχουμε λοιπόν το ζήτημα της συμφωνίας της PNR με τον Καναδά αναθεωρημένη δηλαδή συμφωνία η οποία ακριβώς λαμβάνει υπόψη τα ζητήματα που έθιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εγώ το παραδέχτηκα από μόνος μου ότι πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα κάνει πάντοτε όλα σωστά. Ε, λειτουργούμε λοιπόν στο πλαίσιο ενό συστήματο δικαίου και ε, μα ελέγχετε κι εσεί και ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μα ελέγχει. Και όταν μα ζητάει το δικαστήριο να εξετάσουμε κάτι εκ νέου, ε, αυτό κάνουμε το εξετάζουμε από νέα οπτική γωνία και η συμφωνία PNR με τον Καναδά επανεξετάζεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο και πιστεύουμε ότι ε, ο Καναδάς θα μπορέσει να κυρώσει αυτή τη νέα συμφωνία. Τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως ε, θα γνωρίζετε ξέρετε μάλλον τι συμβαίνει εκεί ενώ με την ε, Αυστραλία έχουμε ξεκινήσει μια πρώτη αξιολόγηση του Εδώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ε, μια τέτοια συμφωνία ειναι μαζί του Εδώ η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ε, ε, έγινε μια συζήτηση καταρχήν με τι ΗΠΑ στην οποία συζήτηση θα δοθεί συζήτηση το Σεπτέμβριο, ενώ τον Αύγουστο θα μεταβούμε και στην Αυστραλία και βέβαια θα συνεχίσουμε να σα ενημερώνουμε σε σχέση με τις διαδικασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, την καλύπτουμε στο πλαίσιο της έκθεσής μας ε, και γνωρίζετε ότι έχουμε εργαστεί σκληρά σε σχέση με αυτή την ε, οδηγία και έχετε δει το τι κάνουμε. Έχουμε 25 κράτη-μέλη τα οποία έχουν μεταφέρει στην εθνική του νομοθεσία αυτή την οδηγία, ενώ υπάρχει ένα κράτο μέλο το οποίο η Σλοβενία συγκεκριμένη που ακόμα δεν έχει μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία αυτή την οδηγία και υπάρχει ένα ακόμα κράτος μέλος το οποίο έχει αναλάβει μεν την δέσμευση να το κάνει, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα με την έγκριση από το Κοινοβούλιο τη εν λόγω ε, οδηγία και αυτή η χώρα είναι η Ισπανία και είχαμε μάλιστα και διμερή επαφή με την Ισπανία ε, χθε. Δεν έχω λοιπόν καμία αμφιβολία ε, ω προ την βούληση αυτών των δύο κρατών μελών να τηρήσουν τα όσα συμφώνησαν, αλλά υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση, ειδικότερα στην Ισπανία σε σχέση με το Κοινοβούλιο και θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα και τα υπόλοιπα, εμεί θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και βέβαια θα του ζητούμε το λογαριασμό, αν θέλετε, εάν ή θα του ζητήσουμε το λογαριασμό, αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που έχουν ε, αναλάβει, στι δεσμεύσει που έχουν αναλάβει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα τη διαλειτουργικότητα και πάλι τις, ε, τα όσα έχουν πει ότι θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολο αυτό το ζήτημα. Το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε ευθύ εξ αρχή όταν είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Πρόκειται δηλαδή για ένα μεγάλο εγχείρημα το να πούμε ότι θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τι βάσει δεδομένων, τι υφιστάμενες και να δημιουργήσουμε κάποιε νέε ε, ε, βάσεις δεδομένων, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το συστημα εισοδου εσόδου-εξόδου, το ETS. Και βέβαια όταν λέμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τη διαλειτουργικότητα με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός μεν, αλλά με όλες τις προστασίες, με όλες τις κλίδες ασφαλείας που αναφέραμε ήδη. Και είπαμε ότι υπάρχει χρηματοδότηση, υπάρχουν κονδύλια από τη δικιά μας ε, πλευρά διαθέσιμα, υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη την οποία θέλουμε να μοιραστούμε με τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε για λογαριασμό των κρατών μελών αυτών. Και το αναφέραμε και σε υπουργικό επίπεδο. Και το κάναμε και τώρα. Την ε, περασμένη εβδομάδα δηλαδή στο άτυπο Συμβούλιο ΔΕ. Και είχαμε και μία σειρά από συζητήσεις με τις αρχές των κρατών μελών, όπου ακριβώς ε, εξετάσαμε τις λεπτομέρειες του πώς θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η πρόταση και αν, σας, ε, αν θέλετε θα συνεχίσω να σας ενημερώνω σε σχέση με το λόγο ζήτημα και το πώς προχωράμε. Πρέπει να σας πω ότι κάναμε μια συνολική αξιολόγηση της ε, υλοποίησης ε, συμπεριλαμβανομένου και του, της πτυχής ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όταν ήρθα εδώ το 2016 στην αρχική μου ακρόαση, το είχαμε ήδη αναφέρει αυτό και ορισμένοι μεταξύ ημών μου ζητήσατε να το κάνω και το κάναμε. Εκατοντάδες είναι οι σελίδες ε, και το δώσαμε το αποτέλεσμα σε αυτήν την Επιτροπή. Ε, λυπούμε εάν δεν το είδατε ε, και αν δεν το καταλάβατε ότι υπάρχει η έκθεση αυτή. Ε, κοιτάξτε, έχουμε 15 χρόνια ε, πρωτοβουλειών στον τομέα αυτό, αλλά πρώτη φορά έγινε αυτή η αξιολόγηση. Αν θέλετε τώρα να το επικαιροποιήσουμε, ε, με μεγάλη χαρά θα το κάνουμε. Όσον αφορά, ένα, κάποια συγκεκριμένα αδύναμα σημεία για την υλοποίηση, έχετε δίκιο όταν υπογραμμίζεται κάποια λεπτομερή στοιχεία ε, για το πακέτο ε, κατά του ξεπλήματος ε, χρήματα. Ναι, δεν έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε. Το συζητήσαμε μάλιστα και σήμερα το πρωί στο κολέγιο των Επιτρόπων όπου είδαμε τρόπους ε, για ενίσχυση της ε, ε, συμφωνίας για το ξέπλυμα χρήματος. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξαναδούμε και να δούμε πώς, πώς ακριβώς φτιάχνουμε αυτήν την νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος. Υπήρξε και μία ερώτηση υπήρξε μία ερώτηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων και την διακράτηση των δεδομένων. Ε, κυρία Στρίκ, ε, μου κάνατε μία ερώτηση η οποία σχετίζεται με το PNR στην ουσία. Συμφωνήσαμε όμως ε, ε, ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις για το θέμα αυτό και με εσά, με τους συνομοθέτες. Υπάρχει όμως ακόμα ένα εκρεμές ερώτημα, δηλαδή πώς θα δούμε στο μέλλον αυτό το θέμα της γενικής διακράτησης ε, των δεδομένων, γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σχήμα γι' αυτό. Ε, εμείς ε, έχουμε συζητήσει με πολλούς εμπειρογνώμονες για τα θέματα αυτά και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και βεβαίως θα αναφερθούμε σε εσά και στο Συμβούλιο για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και το θέμα με τις εκρεμούσες ε, ε, ενώπιον του δικαστηρίου ε, υποθέσεις, γιατί υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις. Τέλος, και ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις, υπήρξε μία ερώτηση για το τράφικινγκ, καθώς επίσης και για την και για την διακίνηση ε, μεταναστών. Ε, ε, υπάρχει ένα καινούριο κέντρο για την αντιμετώπιση ακριβώς της διακίνησης και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι, λέει ο Πρόεδρος, που ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο. Έχουμε τώρα πολλές, πολλούς συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Εάν θέλουμε να μιλήσουν όλοι στο χρόνο που έχουμε, θα πρέπει να μην ξεπερνάει ο καθένας μας το 1,5 λεπτό, έτσι ώστε να υπάρχει και χρόνος για απαντήσεις. Δηλαδή να πάρετε το λόγο, αλλά να μην ξεπεράσετε το 1,5 λεπτό ο καθένας. Now with uh, uh, our Vice Chair, Mr. Radev. Ο κύριος Ράντεφ, 1,5 λεπτό παρακαλώ, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε Κίνγκ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για την εξαιρετική και καρποφόρα συνεργασία που είχαμε ε, στην προηγούμενη θητεία. Κυρίως δεν σας ευχαριστήσω γιατί βελτιώσατε το σύστημα διασυνοριακής πρόσβασης σε αποδεικτικά στοιχεία ε, για τις διοκτικές και άλλες αρχές. Το ζήτημα του ξεπλήματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι έχουν καταχραστεί ε, οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες γενικώ ε, των συστημάτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ε, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Ε, για την ώρα ε, όλα αυτά διέπονται από εθελοντικό χαρακτήρα στα και θα πρέπει οπωσδήποτε να, ε, στην περίπτωση ειδικά των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων να είναι αμφίδρομη η σχέση στις ε, συζητήσεις ε, στα πλαίσια ΔΕΗ που έχετε κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, λέτε ότι πρέπει να υπάρχει ακριβώς αναλογικότητα και αμοιβαιότητα μάλλον μεταξύ των χωρών. Ωστόσο, η χώρα μου η Βουλγαρία έχει πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν ε, να κινηθούν ελεύθερα. Ε, πιστεύετε ότι για τις 7 χώρες οι οποίες ακόμα έχουν υποχρέωση θεώρησης ε, θα αρθεί η υποχρέωση αυτή. Επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις. Ε, το, ανθρώπινο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε ένα κράτος μέλος γιατί δεν ε, ε, φύρμωσε σωστά την νομοθεσία σε μια περίπτωση δολοφονίας τρομοκράτη. Η ηθική ζημία υπήρξε μεγάλη γιατί της οικογένειας του θύματο εννοώ γιατί αυτή η κυρία ζει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς λέτε επίσης ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν τα συστήματα και θα πρέπει και εμείς ε, να ε, ε, προσαρμοστούμε το, στο θέμα των, των, της αναγνώρισης των το, του μηχανισμού αναγνώρισης ε, και των δικαιωμάτων εδώ. Το συζητήσαμε στην, ε, στο Κοινοβούλιο, ε, αλλά όταν έχουμε τόσο πολύ σημαντικές εγκληματικές πράξεις και ποινικέ όπως είναι το, η τρομοκρατία, θα πρέπει να βρούμε έναν ειδικό τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Επίσης, το θέμα των υβριδικών απειλών εδώ. Έχουμε μία πρόταση από πλευράς ε, της, ε, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου που ζητάει να δημιουργηθεί μία σπίδα προστασίας ευρωπαϊκή στον Περσικό κόλπο και το λέει τώρα, λίγο πριν από το Brexit. Brexit. επίσης, όσον αφορά το Γιβραλτάρ, το λάβατε υπόψη σας. Είναι μια ειδική περιοχή η οποία δημιουργεί ε, γύρι προβλήματα. Κυρία Κινίτση, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Κίνγκ και για την εργασία που έχει κάνει μέχρι τώρα όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας, αλλά και για την καλή συνεργασία που είχαμε ε, μεταξύ μας και βεβαίως για αυτόν τον συνεχή διάλογο με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Για όλα αυτά τον ευχαριστώ. Είναι σημαντική η νομοθεσία που παρήχθη στην προηγούμενη ε, θητεία και που ενίσχυσε το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο καθώς επίσης ε, και την συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων ε, στον ποινικό τομέα και όσον αφορά τρομοκρατία και όσον αφορά διακυβερνητικό έγκλημα και ανταλλαγή πληροφοριών για οικονομικά εγκλήματα κλπ όλα τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά για την ε, αντιμετώπιση των ε, διασυνοριακών εγκλημάτων που οργανώνονται ακριβώς από το οργανωμένο έγκλημα. Ελπίζω ότι και τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Αλλά δεν θεωρείτε ότι ακόμα πολλά μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να ενισχυθεί ε, ε, το νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της, ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι πάνω από 5.000 οι οργανωμένες αυτές ομάδες που βέβαια έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους bikers μέχρι το πιο, τις πιο οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει, μάλλον δεν νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να έχουμε ε, μια συγκεκριμένη ε, νομοθεσία ε, που θα αναφέρεται στο ισχύο νομοθετικό πλαίσιο και θα το ενισχύει. Κυρία Στρουγκάρη, παρακαλώ, 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι που σας βλέπω. Ω μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέβαλα στην εργασία για τα θέματα αυτά όταν ήμουν μέλος του προσωπικού. Τώρα είμαι από διαφορετική θέση. Πρώτη ερώτηση. Πείτε μας λίγο περισσότερα για τις προτεραιότητες της επόμενης Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια και τις υβριδικές απειλές. Και δεύτερον, το 5G. Η Κατρίν Ντεμπόλ, που είναι επικεφαλής της Europol την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι οι ευρωπαϊκές αστυνομικέ αρχές δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν και τις συνομιλίε και τις μετακινήσεις των εγκληματιών ε, με το 5G κάτι που είναι δυνατό τώρα με το δίκτυο 4G και οι εφημερίδες ε, αυτό το παρουσίασαν ως ε, θέλετε να είστε εγκληματίας περιμένετε να περάσουμε στο 5G. Μπορείτε να μας πείτε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Μπίσεκ, ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη για την τεχνική δυσχέρεια. Είμαι νέο μέλος και στη Λίμπε και χαίρομαι πολύ που θα μπορούσα να δουλέψω για αυτά τα θέματα. Με ικανοποίησε το ότι μιλήσατε αναλυτικά για το θέμα της παραπληροφόρησης που αντιμετωπίζουμε στην Ένωση. Χαίρομαι που έχει γίνει ουσιώδες θέμα. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή με τις προεκλογικές περιόδους. Είναι καθημερινότητα. Θα πρέπει λοιπόν να είναι ε, καθημερινό μας μέλημα. Αυτό λοιπόν ρωτάω. Πώς θα γίνει η πραγματική πολιτική προτεραιότητα, όχι μόνο για τα θεσμικά όργανα. Τι συστάσεις έχετε για την επόμενη Επιτροπή Και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης ε, μας ενδιαφέρει και από πλευράς ε, σε διάφορα κράτη-μέλη. Προτείνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάτι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ κυρία Ίντσερ. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ήδη έχει τεθεί αλλά με διαφορετική διατύπωση. Η τρομοκρατία είναι τρομοκρατία ανεξάρτητα από την ιδεολογική του τοποθέτηση. Το ένα είναι αντικατοπτρισμός του άλλου, οι τζιχαντιστές και οι ακροδεξιοί. Το 2017 είχατε ήδη ειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή της ακροδεξιάς τρομοκρατίας στην Ευρώπη και είπατε ότι αυτή η ακροδεξιά τρομοκρατία είναι, ένας, ε, είναι μια απειλή ε, η οποία δεν είναι τόσο παρούσα στην, ε, στα μέσα όσο η Ισλαμιστική. Η πολιτική διάσταση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας πολύ συχνά υποτιμάται. Δυστυχώς και από συναδέλφους εδώ και ε, οι τρομοκράτες, οι ακροδεξιοί τρομοκράτες ε, παρουσιάζονται απομονωμένα άτομα και με προβλήματα ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, πριν από 8 χρόνια είχαμε τα άτομα που σκοτώσανε τόσους ε, σε αυτό το νησί έξω από το άτομο που σκότωσε όλα αυτά τα άτομα σε αυτό το νησί έξω από την Νορβηγία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε αν η ακροδεξιά τρομοκρατία είναι τόσο σοβαρή όσο ήταν το 2017 που δώσατε αυτή την απάντηση στο Euroactive και παίρνετε εσείς ως Επιτροπή αρκετά σοβαρά αυτή την απειλή και τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε σε ενωσιακό επίπεδο για να καταπολεμήσουμε αυτή την απειλή. Ευχαριστώ πολύ. Λουαζό. Από το Renew. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε. Ο Μπορί Τζόνσον ε, σήμερα γίνεται πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπε ότι όπως και να είναι 31 Οκτωβρίου θα φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω να κάνει λάθος, αλλά ποια είναι η γνώμη σα. για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσουν μια άτακτη έξοδο, ιδιαίτερα από πλευρά ασφάλειας. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε στη σημασία της κυβερνοασφάλειας για την Ένωση. Ποια είναι η γνώμη σας για το επίπεδο ετοιμότητας των ενωσιακών θεσμών για να αντιμετωπίσουν τέτοιες απειλές. Τι έχουμε κάνει, τι πρέπει ακόμη να κάνουμε. Υπάρχουν προπαρασκευαστικές εργασίες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μάγκιντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση, Επίτροπε Κίνγκ. Λοιπόν, καλωσορίζω την πρόσφατη είδηση ότι οι Βρετανικέ Υπηρεσίε Ασφαλείας αντιμετωπίζουν σοβαρά τον ακροδεξιό κίνδυνο και έχουν ε, αναβαθμίσει το επίπεδο κινδύνου. Αλλά λόγω της ε, φρικόδους δολοφονίας ε, της βουλευτού Joe Kicks, από έναν ακροδεξιό τρομοκράτη, λόγω των επιθέσεων κατά τον Ρωμά και των επιθέσεων άλλων που πιστεύουν στην ανωτερότητα της λευκής φυλής παντού στην Αφρική και ο Καναδάς επίσης έχει ε, αναβαθμίσει το επίπεδο απειλής από αυτούς. Λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτοί οι οπαδοί της ε, ανωτερότητας της λευκής φυλής ε, αντιμετωπίζονται σοβαρά με, τις, με τους κατάλληλους πόρους και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι θα προτείνετε στο διάδοχό σας για να βελτιωθεί η αντιμετώπιση. Ευχαριστώ κυρία Στάντλερ. Ευχαριστώ. Καλώ ήρθατε κύριε Επιτροπέ. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπω. Επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ελπίζω να μην γίνει Brexit και να είστε εδώ και στην επόμενη θητεία. Οι παρατηρήσει σα δείχνουν ότι η ασφάλεια είναι πολύ ευρύ τομέα. Συμφωνούμε με αυτό που είπατε, ότι από κοινού μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Είναι πολύ απαιτητικό ο αλλά είναι και βασική ανάγκη σε όλε τι κοινωνίες. Υπάρχουν προφανείς απειλές όπως τρομοκρατία, αλλά υπάρχουν και άλλες απειλέ. Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις, τις αναφέρατε. Υπάρχουν οι κρίσιμε ψηφιακέ υποδομές. Αλλά ας αφήσουμε τη λέξη ψηφιακή. Τώρα πια όλες οι υποδομές είναι με τον αβ τρόπο ψηφιακέ. Οπότε, πόσο καλά έχουν προετοιμαστεί για τη χειρότερη εναλλακτική λύση, για παράδειγμα σοβαρέ διακοπές ρεύματο. Και δεύτερο θέμα, η Europol. Θαυμάσια δουλειά κάνει. Έχει ευρύ πεδίο δραστηριότητα ιδιαίτερα... Συγγνώμη, έχει ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, αλλά δεν έχει επαρκεί πόρους, ούτε επαρκέ προσωπικό. Και υπόθηκε ότι θα περικοπούν 52 θέσεις ε, ορισμένης διάρκειας και 33,7 εκατομμύρια από τον προπολογισμό της. Τι νομίζετε εσείς για αυτά τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, Europol. Πρέπει να της δώσουμε όλα όσα θέλει και για τον τρόπο λειτουργίας και για τους πόρους και το προσωπικό. Ε, ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, για την παρουσίασή σα ε, και υπάρχουν πολλά τα οποία έγιναν από πλευρά τη Επιτροπή και θα ήθελα να σα ευχαριστήσω προσωπικά για το γεγονό ότι έχετε πραγματικά αφοσιωθεί στην ε, κυβερνοασφάλεια. Περνάμε δύσκολου καιρού δηλαδή. βλέπουμε τι συμβαίνει με τι τεχνολογίε πληροφορική και το γεγονό ότι οι κυβερνοεπιθέσει αποτελούν μια πραγματικότητα σήμερα. Υπάρχει και ιδεολογικό χάσμα σήμερα στον κόσμο και έτσι αυτό απηχείται και στην, στα ζητήματα τη κυβερνοασφάλεια. Υπάρχουν ζητήματα επίση εφαρμοσιμότητα του διεθνού δικαίου παρότι έχουμε τηρήσει αυστηρή στάση από την πλευρά μα. Οπότε, μέσα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, ποιο ρόλο θεωρείτε πω μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την εφαρμογή της διεθνούς, του διεθνού δικαίου και πώ μπορούμε να ε, ενισχύσουμε περισσότερο τη διεθνή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως βασικό παίκτη ε, για την βελτίωση της ε, ανταπόκρισής μας σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Ο ε, ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, διάβασα τα όσα έχετε δημοσιεύσει και άκουσα τα όσα είπατε τώρα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα κυβερνού ασφάλεια. Συμφωνώ μαζί σα και θα ήθελα να θέσω δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, ω ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο, εμεί ε, δεν ακολουθούμε κατά πόδος ε, τα όσα συμβαίνουν στο επίπεδο κυβερνού ασφάλεια τη ΗΠΑ και την Κίνα σε ό,τι αφορά αυτές τις απειλές. Και βέβαια θα πρέπει να αναπληρώσουμε αυτό το ε, κενό όχι μόνο για οικονομικά συμφέροντα, ακριβώς, ε, αλλά ακριβώ επειδή υπάρχουν ευάλωτα σημεία. Ε, και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, και τα συστήματα λογισμικού, υπάρχουν κάποια μονοπόλια εδώ, κάποιε εταιρείε δηλαδή που έχουν το μονοπόλιο και οι οποίε δεν εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτέ οι εταιρείε και αυτά τα λογισμικά συστήματα βρίσκονται στην καρδιά των συστημάτων πληροφορική μα. Οπότε αυτό ίσως θα πρέπει να το ε, να το κληροδοτήσετε στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ε, το να αντιμετωπιστούν αυτά τα τεχνολογικά ζητήματα που έχουμε. Ένα δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι τα ζητήματα ηθικής σε σχέση με την τεχνολογία. Νομίζω πως ε, είναι προς το συμφέρον μας να διατηρήσουμε τον τρόπο ζωή μας ο οποίο ο τρόπο ζωή μα επηρεάζεται όλο και περισσότερο από αναλλακτικέ μορφέ διακυβέρνηση και αναλλακτικέ αρχιτεκτονικέ στον ε, online κόσμο. Οπότε, όσο το δυνατόν εμ, αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το πώ θα εντυπώσουμε ακριβώ ε, σε αυτού του τομεί την δική μα τι δικέ μα αρχέ, για παράδειγμα και στη τεχνική νοημοσύνη, τόσο πιο ευπρόσδεκτε θα είναι αυτέ οι νέε τεχνολογίε μέσα στι ε, ζωέ μα. Νομίζω λοιπόν πω αυτά τα δύο ζητήματα θα πρέπει να μα απασχολήσουν στο μέλλον. Ευχαριστώ, πρώτο, κύριε Μπάρλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ στι εξαρτήσει παραπληροφόρηση τι οποίε αναφέρατε, κύριε Επίτροπε, ε, και συμμεριζόμαστε την άποψή σα ότι δεν ήταν τόσο ε, ε μεγάλος ο αρνητικό αντίκτυπος τέτοιων επιθέσεων στο πλαίσιο των ευρωεκλογών μα όσο αυτούς που φοβόμασταν. Και σε σχέση με αυτό θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέποντα τα πράγματα λίγο αναδρομικά, θεωρείτε πω ε, κάναμε πράγματι αρκετά από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή απλά ήμασταν τυχεροί. Και τα κράτη-μέλη είναι προετοιμασμένα για τέτοιου είδου εξαρτήσει παραπληροφόρηση, οι οποίε θα. με τι οποίε θα βρεθούν αντιμέτωπα τα κράτη-μέλη και στο μέλλον. Και το τρίτο ερώτημα που είχα ήδη έχει τεθεί από τον συνάδελφο σε σχέση δηλαδή με το αν θα υπάρξει νομοθεσία σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, και μάλιστα σας θυμόμαστε παλιότερα ως πρέσβη της χώρας σας στην ε, Γαλλία και εκεί είσαστε ιδιαίτερα ε, ενεργητικός ότι μείνετε λίγους μήνες μόνο. Ερώτηση. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά τη μείωση του προσωπικού της Europol που προβλέπεται στον προϋπολογισμό 2020 και που ε, αντιπροσωπεύει μείωση 25% περίπου. Ε, το, η Ευρωπόλ ε, είναι στο σύστημα, το σύστημα EIS και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση ε, υπόπτων. Επίσης, ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την παρακολούθηση των οικογενειών που επιστρέφουν από τις ε, του πολέμου. Κυρία Μπλίξ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε, κύριε Επίτροπε, σε το, στην προβληματική των ε, ε, ξένων ε, μαχητών και την υποστήριξη δράσεων όσον αφορά κυρίως τον επαναπατρισμό τους, αλλά κυρίως των παιδιών αυτών που βρίσκονται Συρία, στη Συρία και στο Ιράκ. Βεβαίως επίγει η κατάσταση από ανθρωπιστικής απόψεως, κυρίως γιατί τώρα έχουμε πολύ ζέστη και σίγουρα θα έχουμε θανάτους λόγω της ζέστης, ακριβώς όπως είχαμε άλλωστε και θανάτους και ε, λόγω του ψύχου στο χειμώνα. Μην λησμονούμε ότι 90% ε, των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτά τα στρατόπεδα, στις χώρες αυτές, 90% λέω είναι γυναίκες και παιδιά. Δεύτερη κατεπίκουσα κατάσταση ε, είναι αυτή η οποία αφορά την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και κάθε μέρα που περνάνε εκεί τα παιδιά ε, τόσο περισσότερο ε, υφίστανται την, ε, την επίδραση των διδαχών ας πούμε των τζιχαντιστών. Θα πρέπει οπωσδήποτε και να τους δώσουμε την δυνατότητα τα παιδιά κυρίως να ζήσουν αξιοπρεπώς, να ζήσουν σαν παιδιά και να τους δώσουμε και την δυνατότητα να έχουν ένα μέλλον. Βεβαίως όπως και το είπατε άλλωστε αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά από τη στιγμή που το θέμα αυτό μπορεί να ενταχθεί ή στην γενικότερη αντιμετώπιση της τρομοκρατίας θα μπορούσε να περάσει και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, με μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύρια. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φέστα Ιντύπ. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών είναι η βάση της δημοκρατίας. Και αυτό το βλέπουμε σε δύο περιπτώσεις. 25 Μαΐου στη Λιόν έγινε μια τρομακτική επίθεση του Ισλανδικού, του Ισλαμικού κράτους. Και το κάλυψε η κυβέρνηση Μακρόν. Και αυτό έπαιξε ρόλο στη σύσταση αυτής τη Επιτροπής. Το ότι δεν το έκανε γνωστό. Επίσης, ε, στο γερμανικό στρατό υπόθηκε ότι υπάρχει ένα ακροδεξιό δίκτυο, αλλά δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, γιατί ορισμένε ε, ε, έρευνε ούτε καν ξεκίνησαν λόγω, λόγω του δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία καταλαβαίνετε τι σημασία έχει να ασχοληθείτε και με αυτές τις υποθέσεις. Τι αξιοπιστία έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η πρόεδρος του ω Υπουργό Άμυνα συμμετείχε σε αυτήν την εκστρατεία παραπληροφόρηση του γερμανικού κοινού. Ο κύριος Αλσαλάνη, η κυρία Αλσαλάνη από το Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πολλά μας είπατε. Κύριε Επίτροπε, μια ομάδα για την οποία μιλάμε πολύ λίγο όταν μιλάμε για την προστασία των συμπολιτών μας από τρομοκρατικές επιθέσεις είναι τα άτομα που δρούν με τρόπο συγγνώμη η δραστηριότητά τους ε, του, τους κάνει πολύ εκτεθειμένους σε επιθέσεις. Αλλά η οδηγία δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Αλλά θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες αυτών των ατόμων. Εάν δεν υπάρχουν ε, μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρότεινα το θέμα αυτό να είναι προτεραιότητα γιατί αφορά την ασφάλεια όλων μας. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι πρέπει να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ατόμων στις νέες προτάσεις πολιτικής που κάνετε για την ασφάλεια. Ο, ο κύριος Παπαδάκης, 1,5 λεπτό. Ε, τι μας είπατε εδώ, ότι πρόταση λέγεται μαζικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων και κάποτε στο μέλλον θα φτιάξετε ένα πλαίσιο διατήρησης αυτών των δεδομένων. Οι δημοκρατικές ελευθερίες και τα δικαιώματα δηλαδή βρίσκονται στο στόχαστρο και εσείς επιχειρείτε να ξεμπερδέψετε με ευχές για προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή για το JDPR. Ποιο άραγε μπορεί να ελέγξει για το τι και πώ συλλέγεται στο όνομα τη ασφάλεια, Ποιο να ελέγξει του μηχανισμού, του πολυπλόκαμου, το δίκτυο παρακολούθηση, τη δακτυλοσκόπηση, τη συγκέντρωση δεδομένων πληροφοριών με επεξεργασία στοιχείων σε διασύνδεση με μεγάλου ομίλους τηλεπικοινωνιών με πώληση ή διαρροή στοιχείων για εμπορικούς ή πολιτικούς λόγους. Σήμερα οι λαοί είναι εκτεθειμένοι από την καταγραφή από το απλό κλικ στο κομπιούτερ τους μέχρι την ενοχοποίησή τους ακόμα και για ταξιδιωτικούς προορισμούς. Ριζοσπαστικοποίηση λέτε, έννοια που με αυθαίρετο τρόπο γίνεται λάστιχο, ενοχοποιείται η συμμετοχή στο εργατικό κίνημα, η συνδικαλιστική δράση, διώκεται ακόμα και απλή απεργία τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί άνθρωποι με υποψίες και αυθαίρετες ερμηνείες. Αλήθεια, πού ξεκινά και πού σταματάει η ριζοσπαστικοποίηση. σκοπι θολούρα. Άλλωστε, ξέρετε καλά ότι οι γνωστές ομάδες για την αποκρουστική δράση τους είναι γνωστό ότι χρηματοδοτήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν από τις ΗΠΑ, από κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές οι ομάδες έγιναν πιόνια σε ανταγωνισμούς και πολέμους. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο θα μα προστατέψει από του προστάτε. Είμαστε βέβαιοι ότι οι λαοί θα σπάσουν τι αλυσίδε του και τι ηλεκτρονικέ που του φοράτε αυτή την περίοδο. Mr. Rangel. Ε, uh, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε κάποια διαφορετικά σημαντικά ζητήματα. Καταρχήν, η αντοχή ε, σε επιθέσεις και ασφάλεια των ε, δικτύων 5G. Ε, μας είπατε ότι πρόσφατα τα κράτη-μέλη έχουν παρουσιάσει και έχουν ολοκληρώσει τις εθνικές τους αξιολογήσεις. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω. Οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, όπως θα γνωρίζετε, έχουν θέσει αμφιβόλω την αξιοπιστία των δικτύων 5G, ειδικότερα των ε, ευρυτά ευρυζωνικά. Τα ε, ειδικότερα της εταιρείας Huawei. Ε, δηλαδή υπάρχουν κάποιες ε, υποψίες σε ό,τι αφορά την χρήση από την Huawei αυτών των δικτύων 5G ε, για το mining δεδομένων, δηλαδή τη συλλογή δεδομένων. Έχει κάνει κάποια σκέψη σχετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το λαμβάνει υπόψη στο πλαίσιο της σύναψης συμφωνιών στον τομέα της ασφάλειας. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά τα συστήματα πληροφορικής. Όπως ε, θα γνωρίζετε από την προηγούμενη βουλευτική θητεία, εγκρίναμε την οδηγία της καταστάσεων ομάδων ε, επιβατών, την PNR. Έχω αντιληφθεί σωστά το ότι ε, διενεργείται αυτή την περίοδο ένα πιλωτικό project του, ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή αυτή τη οδηγία σε PNR. Και αν ισχύει αυτό, μπορείτε να μα πείτε δύο για παραπάνω. Κύριο Κόνορ, τώρα από το Renew Europe. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Επίτροπο Κίνγκ. Θα ήθελα να θέσω κι εγώ ένα συμπληρωματικό ερώτημα σε σχέση με την οδηγία PNR. Ε, ακούσαμε δηλαδή ότι υπάρχουν αξιολογήσεις αυτή την περίοδο από τα κράτη-μέλη. Ε, και ε, σε ό,τι αφορά την χρήση τους και για τα άλλα είδη μεταφορών, δηλαδή τη χρήση τους και σε λεωφορεία, στο σιδηρόδρομο, ακόμα και σε ε, πλοία, τι σκέφτεστε. Ε, στη Γερμανία και ήδη από τον συνάδελφο το 99,7 των hits, των θετικών δηλαδή αποκρίσεων μέσα στο σύστημα, είναι σφαλμένα, είναι, είναι ψευδείς ε, θετικές αποκρίσεις. Και είδαμε ε, και τι ε, φρικτέ επιθέσεις όταν αφορά την αξιοπρέπεια των ε, ατόμων από τον τομέα LGBTI, στην, των ΛΟΑΔΜ δηλαδή, στην Πολωνία. Πώς μπορείτε λοιπόν να παράσχετε προστασία σε αυτά τα άτομα από την κατάχρηση αυτού του συστήματος. Ευχαριστώ. Λέω, ο Πρόεδρος, έχουμε ξεπεράσει και πάλι αυτό το, το, το τα χρονικά μα πλαίσια εδώ και ευχαριστούμε εκ των προτέρων τους διερμηνείς μας που θα παραμείνουν για 15 λεπτά ακόμα ε, μαζί μας ε, και αυτό γιατί αυτό το ζήτημα γενικότερα της στρατηγικής ασφάλειας μας απασχολεί πάντοτε και ε, γι' αυτό όμως θα ήθελα να παρακαλέσω και τους υπόλοιπους ομιλητές πραγματικά να τηρήσουν εδώ τα χρονικά τους όρια του χρόνου αγόρευσης δηλαδή ώστε να έχετε δυνατότητα και ο Επίτροπος να απαντήσει. Ο κύριος Ζεμπράιερ έχει τώρα το λόγο από τους Πράσινους. Ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, είμαι νέο μέλος εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, ε, και έχω περιοριστεί στα βασικά μου ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ζήτημα της συλλογή των δεδομένων στο πλαίσιο της οδηγία PNA, DFTP και την δυνατότητα επέκτασης σε λεωφορεία και σε τρένα, τέτοιου είδους προτάσει έχουν κηρυχθεί άκυρες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ε, Δανία υπήρξαν μια σειρά από υποθέσεις όπου υπήρξαν καταδίκες δηλαδή επί τη βάση ψευδών στοιχείων. Οπότε πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επεκτείνει τώρα τέτοιου είδους πολιτικές ή ε, θέλει να εφαρμόσει πλέον, θεωρεί ότι έχει φτάσει η χρονική ε, στιγμή να τεθεί ένα μορατόριο, να σταματήσουν δηλαδή αυτά τα προγράμματα μαζικής ε, παρακολούθηση μαζική ε, συλλογή δεδομένων. Τώρα, σε ό,τι αφορά ειδικότερα το ζήτημα τη οδηγία PNR, καθώ το δικοστήριο έχει θεωρήσει πω η συγκεκριμένη πολιτική είναι δυσανάλογη, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν οδηγεί ενώπιον του δικαστηρίου τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν ε, τηρούν το σχετικό περιορισμό και συνεχίζουν δηλαδή να εφαρμόζουν με αυτόν τον τρόπο την οδηγία PNR. Τέλο, σε ό,τι αφορά το ζήτημα ε, του τρομοκρατικού περιεχομένου online, έχετε στη διάθεσή σα σαφή αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να καταδεικνύουν ότι η διαγραφή τρομοκρατικού περιεχομένου online μειώνει την τρομοκρατία. Ε, δηλαδή, έχετε κάποια πραγματικά στοιχεία αξιόπιστα που το καταδεικνύουν αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, ο κύριος Γκαρό τώρα από το ID. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, αναφέρατε ότι θέλετε να ε, απαντήσετε με ασφάλεια ε, στο, στην ριζοσπαστικοποίηση και στο αφήγημα μίσους επιγραμμικά. Όσον αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση, υπάρχει ένας τόπος που πραγματικά υπάρχει μεγάλος βαθμός ριζοσπαστικοποίησης. Είναι τα σοφρονιστικά ιδρύματα. Θα πρέπει να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο στο θέμα αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά την, το κυβερνοέγκλημα, είπατε ότι έπρεπε να, πρέπει να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρέσουν το περιεχόμενο τρομοκρατικού περιεχομένου, τρομοκρατικών ε, site. Αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος. Μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ποινικοποιήσουν ε, το, αυτού του είδους το περιεχόμενο. Ε, θα πρέπει να ποινικοποιηθούν σε όλες τις χώρες ε, τα περιεχόμενα, τα τρομοκρατικά περιεχόμενα. Τέλος, όσον αφορά το, τον λόγο μίσους, ο λόγος μίσους ξέρουμε τι σημαίνει. Αναφερόμαστε σε παρακίνηση στην βία, ε, αυτό είναι σαφές, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Ε, υπήρξε ένας πρώτος νόμος κατά κάποιο ε, τρόπο στον λόγο μίσους στη Σοβιετική Ρωσία. Δεν χρειάζεται βέβαια να φτάσει μέχρι τις, τους αντιφρονούντες. Θεώρησα ότι μέχρι εκεί θα μπορούσε να φτάσει ο λόγος μίσους, το να εκφράσει δηλαδή κανείς μια διαφορετική γραμμή από την κυβερνητική. Να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Yes, please. Thank you. Okay. Ευχαριστώ. Πρώτον, ακραίο περιεχόμενο στη, στη μέσα κοινωνική δικτύωση. Πολύ σημαντικό. αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να παριλάβετε μόνο την άμεση παρακίνηση σε, για, σε βία. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι με του οποίου θα μπορούσατε να παρακινήσετε προ αυτήν την κατεύθυνση. Το Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ακροδεξιοί ακτιβιστέ δημοσιεύουν περιεχόμενο που μπορεί να υπονομεύσουν τις δίκαιε δίκε. Ξέρετε ότι υπάρχει κάποιο που λέγεται Τόμι Ρόμπινσον που ε, ε, φυλακίστηκε για τέτοια πράγματα 9 μήνες και δεν είναι ο μόνος. Μπορείτε να εξετάσετε και τέτοιου τύπου συμπεριφορά λοιπόν να τη συμπεριλάβετε. Και μια σοβαρή απειλή σε πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρε είναι τα εγκλήματα με μαχαίρια που σκοτώνει πολύ περισσότερο άτομα τον χρόνο από την τρομοκρατία. 17.500 14χρονων αποκάλυψε μία έρευνα στον Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επάνω τους μαχαίρια τακτικά και η κατάσταση με τα εγκλήματα με μαχαίρια στον Ηνωμένο Βασίλειο είναι παράλληλη με την κατάσταση των εγκλημάτων με πυροβόλα όπλα στο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι εύκολο να βουτήξεις ένα μαχαίρι από ένα σούπερ μάρκετ χωρίς να σε πάρει κανείς είδηση και εύκολα μπορείς να αγοράσεις και το διαδίκτυο. Δεν μπορώ να αγοράσω ένα αυτόματο όπλο στη χώρα μου. Γιατί μπορώ να αγοράσω ένα μαχαίρι κυνηγίου ή ένα ε, στρατιωτικό μαχαίρι τόσο εύκολα. Θα πρέπει να τα κοιτάξει αυτά η Ευρωπαϊκή Κέντρο. Ο Μπέργκ, IND. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε Κίνγκ. Η κυβερνοεγκληματικότητα είναι πολύ δυναμική εγκληματικότητα. ω ομάδα, οποιαδήποτε μείωση του προπολογισμού που ε, επιχειρείται από την αριστερά για τις ε, εθνικές αστυνομικέ αρχές για την Europol μας βρίσκουν εντελώ αντίθετους και μας ανησυχούν. Οπότε, τι συστάσεις θα κάνετε στο διάδοχό σας για, ε, για το κυβερνό έγκλημα και σε ποιους τομείς του ποινικού κώδικα θεωρείτε ότι έχουν υπάρξει επιτυχίες για την κυβερνοεγκληματικότητα. Η κυρία Ζίπελ, ε, κάτι πολύ σύντομο πριν επανέλθει ο Επίτροπος Κίνγκ. Ναι, κοιτάξτε. Δεν θέλω πάλι να μου στείλετε τον κατάλογο που, τον οποίο στείλατε όταν μιλήσατε την έκθεση πρώτα από το 2016 γιατί ήταν απλώς οι νόμοι που λέγανε ε, τι ακριβώς κάνει ο κάθε νόμος. Ε, νομίζω ότι ξέρει πολύ καλά ο Επίτροπο Κίνγκ ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι εκθέσει πιο σε βάθο που να δείχνουν πόσο ο συνδυασμό όλων των νόμων και μέτρων θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρω ότι η Επιτροπή ετοιμάζεται τέτοιε εκθέσει, αλλά προ το παρόν ε, δεν έχει καταλήξει η εκπόνησή τη. Ε, δεν ξέρω, ίσω πρέπει να επανέλθετε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, και με τα 15 λεπτά Ίσως να έχουμε πρόβλημα για να ακούσουμε όλες τις απαντήσεις του Επιτρόπου Κίνγκ. Λοιπόν, λοιπόν ε, από τις 16 και 45 και μετά θα έχουμε μόνο αγγλικά. Κοιτάξτε, έγιναν πολλές ερωτήσεις για το κύβερνο έγκλημα και τα ηλεκτρονικά στοιχεία. Αυτά τα θέματα σίγουρα θα συζητηθούν τους επόμενους μήνες και χρόνια. Για το κύβερνο έγκλημα το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Κομισιόν να διαπραγματευτεί την ένταξη σε ένα πρωτόκολλο για το κύβερνο έγκλημα, την σύμβαση για το κύβερνο έγκλημα, που μπορεί βέβαια να επικαλύπτεται με κάποια άλλα εγχειρήματα του Κοινοβουλίου. Τι θα κάνετε ούτως ώστε, ούτως ώστε να μπορέσουν να ληφθούν ε, υπόψη τα αιτήματα του Κοινοβουλίου σε αυτήν την διαπραγμάτευση για ένταξη αυτό το πρωτόκολλο. Παρακαλώ. Είναι πολύ καλό που έρχονται οι επίτροποι σε εμά. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε χρόνο να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα αναλυτικά, αλλά ε, εάν δεν μπορέσετε, παρακαλώ δώστε μας ε, ε εκ των υστέρων κάποιες γραπτές απαντήσεις στα θέματα που ετέθησαν. Καλά, σίγουρα δεν θα μπορέσω να απαντήσω ε, με κάθε λεπτομέρεια όπως θα άξιζε η κάθε ερώτηση, αλλά μπορούμε να έχουμε κάτι δύο συζητήσει. Η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή και για κάποια θέματα, κάπως πιο οριζόντια, μπορώ να σας στείλω και γραπτή απάντηση. Για την κυρία Ζήπελα, εγώ δεν γνωρίζω κάποια έκθεση η οποία να μην έχει ολοκληρωθεί γιατί κάπου την έχουμε μπλοκάρει, αλλά θα ελέγξω. Αν μπορούμε να βελτιώσουμε το διάλογο που έχουμε μαζί σας για την επίπτωση της δουλειά μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, βεβαίω. Ευχαρίστω να το κάνουν. Πολλέ ερωτήσεις για την επόμενη Επιτροπή. Κοιτάξτε, έχουμε τώρα την ε, εκλεγήσα πρόεδρο, θα εκπονήσει την πολιτική της με βάση τις καθημερινές γραμμές που ήδη ανακοίνωσε, δεν πρόκειται εγώ να τις δέσω τα χέρια. Όταν λοιπόν μιλάω για μελλοντικέ εργασίε, σα δίνω απλώ τη γνώμη μου με βάση την πείρα μου, που δεν ξέρω τώρα πώ θα είναι σχετική με, την, ε, με τι αναλυτικέ αρμοδιότητε του κάθε επιτρόπου. Με μια γενική λοιπόν τέτοια προειδοποίηση, τέτοια, σαν αυτέ που έχουν πάνω στα πακέτα, περνάω τώρα σε επιμέρου απαντήσει. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για την αντιμετώπιση τη παραπληροφόρηση είναι πραγματικό κίνδυνο, πραγματική απειλή ασφάλεια, σε παραπληροφόρηση για τι κοινωνίε μα. Για τον τρόπο που κάνουμε την πολιτική μα συζήτηση ή τι πολιτικέ διοργανώσει όπω είναι οι εκλογέ ή τα δημοψηφίσματα και για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε μαζί ω κοινότητε. Γιατί πολλοί από αυτή την παραπληροφόρηση προσπαθεί με τον ΑΒ τρόπο να μα διχάσει. Εσ εμένα υπονομεύει αυτό το κοινό τρόπο ζωής μας. Έχουμε κάνει λοιπόν, θεωρώ, ορισμένα σημαντικά πράγματα και ήμασταν και τυχεροί σε άλλες περιπτώσεις, αλλά σίγουρα δεν αρκούν αυτά που κάναμε. Ελπίζω ότι η Μελλοντική Επιτροπή θα θελήσει να κάνει περισσότερα. Με βάση αυτά που έχουμε ήδη κάνει βεβαίως, αναπτύσσοντας τα περαιτέρω και συγκεκριμένα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τον κώδικα διοντολογίας με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά και το έχω πει και στο παρελθόν, γιατί όχι να δούμε και κάποια μορφή ρυθμιστικών κανόνων. Όχι βέβαια ε, προσπαθώντας να λογοκρίνουμε πολιτικά μηνύματα, δεν θα κρίνουμε εμείς αν είναι κάτι σωστό ή λάθος, αλλά να υπάρξουν μερικοί θεμελιώδεις κανόνες για λόγους διαφάνειας, για παράδειγμα, για θέματα διαφάνειας, για το τι είναι και τι είναι πολιτική διαφήμιση, για το τι κάνουν τα bot, και πώς θα είναι δυνατόν εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητοι, να μπορούν να δουν τι γίνεται με αυτά που δημοσιεύονται. Ελπίζω να κάνουμε περισσότερα για το θέμα αυτό στο μέλλον. Το ίδιο και για γενικότερα τον κυβερνοχώρο. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μερικά πολύ σκόπιμα πρώτα αλλά πάρα πολλή δουλειά έχουμε ακόμη να κάνουμε για την κυβερνοασφάλεια. Κάτι που μας λείπει ακόμη και το οποίο νομίζω το εξετάζει η Επιτροπή ΙΝΤΑ. Η δημιουργία ενός δικτύου κέντρων εμ, αριστείας για τον κυβερνοχώρο για να δούμε με τι πρέπει να ασχοληθούμε. Να ενισχύσουμε επίσης τη διεθνή συνεργασία για την εφαρμογή και του διεθνούς νόμου γι' αυτό ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι στην πρωτοπορία αυτών των θεμάτων. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι. Έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα θέματα αυτά, την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε. Που δεν είναι ταυτόσιμη από κάθε άποψη με την αμερικανική προσέγγιση και είναι πολύ διαφορετική από την κινέζικη. Θα πρέπει λοιπόν να παρουσιάσουμε, να προωθήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε για τη δική μας προσέγγιση. Ιδιαίτερα για το 5G, για το 5G, που είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα. Πρέπει με το τέλος του χρόνου να καταλήξει αυτή η διαδικασία. Α, έφυγε ο κύριος. Αλλά ε, εθνικές αξιολογήσεις έχουν μόλις υποβληθεί από 27 από τα 28 κράτη-μέλη. Αυτές θα τις συνδυάσουμε σε μια ενωσιακή αξιολόγηση των κινδύνων και των σημείων ε, των τροτών σημείων των δικτύων 5G και θα κάνουμε μερικές προτάσεις μέχρι το τέλος του χρόνου για να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό και θέλω να το πω από την πρόκληση της πρόσβασης των αστυνομιών και τον κίνδυνο που λέγεται ότι ορισμένε φορές αντιμετωπίζουμε έναν τοίχο μπροστά μας, το σκοτάδι, όταν ψάχνουμε για πληροφορίες. Υπάρχουν πολλές τεχνολογικές αλλαγές, δεν είναι μόνο το 5G η χρήση της κωδικοποίησης, για παράδειγμα, της, κρυπτογράφηση ε, κρυπτογράφησης καλύτερα. Εκεί πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε μετά από άδεια την πρόσβαση των αστυνομικών αρχών που ψάχνουν, ψάχνουν για στοιχεία κάνοντας τη δουλειά τους, τις ερευνές τους. Πρέπει κάτι να κάνουμε στα πλαίσια της νόμιμης εργασίας αυτών των αρχών. Από την άλλη μεριά βέβαια πρέπει να προστατεύσουμε την υποδομή 5G από μη εγκεκριμένε ε, απόπειρε πρόσβασης, από παράνομους ή ε, κακούς γενικά φορείς που προσπαθούν να μας βλάψουν παρεβαίνοντας στην ψηφιακή μας υποδομή. Και τα δύο θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι και χωρισμένα. Τώρα, πόση σημασία πρέπει να αποδώσουμε στην ακροδεξιά δράση. Επιθέσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΚΙ ή άλλων τμήματων των κοινωνιών μας. Από το 2017, ε, τουλάχιστον από τότε, έχουμε εστιάσει στο θέμα αυτό. Όλα αυτά έγιναν πολύ σαφή νομίζω από την ε, αποτρόπαια δολοφονία της Τζο Κόξ και πρόσφατα στη Γερμανία. Ο κύριος Λούπκε φαίνεται ότι ε, ήταν θύμα ακροδεξιάς τρομοκρατικής επίθεσης. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τα κράτη-μέλη όλα τα αντιμετωπίζουν σοβαρά, δεν το ξέρω, το ελπίζω, αλλά είναι τμήμα της δουλειάς μας να τονίσουμε ότι ναι μεν μας ανησυχεί η συνεχόμενη απειλή από την Ισλαμιστική τρομοκρατία, αλλά παράλληλα ανησυχούμε λόγω άλλων μορφών τρομοκρατίας συμπεριλαμβάνωμένη και της ακροδεξιάς. Τέλος. Για το θέμα των εγκλημάτων με μαχαίρια. Προφανώς. Είναι εγκληματική δραστηριότητα. Μπορεί να οδηγήσει σε τραγωδίες. Θέλουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξουν περισσότεροι έλεγχοι για να μην υπάρχει πρόσβαση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, πυροβόλα όπλα. Είναι βέβαια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά αν θέλετε να το συζητήσουμε, ας το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη. Για το θέμα της ε, Europol. Πολύ το θέσατε. Όχι, δεν προτείνεται περικοπή του προπολογισμού της από ό,τι ξέρω. Υπάρχει πρόταση αύξησης του προπολογισμού αλλά υπάρχει συζήτηση για το εάν επαρκεί αυτή η αύξηση του προπολογισμού. Δεν το ίδιο με περικοπή. Σίγουρα θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Η Europol έχει πολύ σημαντική δουλειά να κάνει και όλο και αυξανόμενη και αυξανόμενη και η σημασία της. Πάντα τη στήριξα όσο μπορούσα. Και έτσι θα προσεγγίσω και οποιαδήποτε συζήτηση του προβλήσμου. Λοιπόν, δύο υποσημειώσει πέρα από το βασικό προπολογισμό της Europol πρέπει να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την Europol να έχει πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Ιδιαίτερα ε, για την αντιμετώπιση των κυβερνοπροκλήσεων υπάρχουν άλλες εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης. Και εδώ και σε άλλες αρμόδιες επιτροπές πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την Europol να αξιοποιήσει αυτούς τους άλλους πόρους. Και τελευταία υποσημείωση. Έχει γίνει συζήτηση για το προσωπικό της Europol. Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν είχαν προσληφθεί ε, με τήρηση όλων των διατάξεων. Πρέπει να δούμε πώς θα το εντοπίσουμε αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να στηρίξουμε την Europol. Για τους ξένους ε, τρομοκράτες μαχητές πολλές ερωτήσεις έκαναν κάποια, κάποιο είδου διασύνδεση ανάμεσα ε, στην ριζοσπαστικοποίηση, τρομοκρατία και ε, μετανάστευση. Uh, but I it. Uh... Ε, ζητούμε συγγνώμη, αλλά η διαρμηνία πρέπει να σταματήσει τώρα. Ευχαριστώ. Between the challenges which undoubtedly exist relating to migration on the one hand and security challenges